Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση, διότι είναι 9 και 3 λεπτά και εντάξει. Πρώτο σημείο στην ημερησία διάταξη είναι η έγκριση αυτής, την οποία έχετε στα χέρια σα. Υπάρχει μια επιθυμία για αλλαγή για τα σημεία 4 και 5. Μερκοσούρ, και κατάσταση πρόοδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων το 4 αλλάξει με το 5 δηλαδή. Άμυνα κατά τον εισαγωγό να γίνει το 4-5 και το 5-4. Αν δεν διαφωνεί κανείς ή δεν έχει άλλες επιδεικνύες, ούτως αποφασίζεται. Και προχωρούμε. Σημείο 2. Ανακοινώσεις κανεί η δεν εχει αλλε επιδεικνυες ουτω αποφασιζεται και προχωρουμε σημειο 2 ανακοινώσει του προεδρου οσοι ηθιστε επειδη ειμαστε παντα παρα πολυ διαφανεί και κρυσταλλινοι μεταδιδεται και αυτη η συνεδριαση στο διαδίκτυο απευθείας και καλώς ορίζω όλους τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες από το Ελσίνκι μέχρι τη Θεσσαλονίκη παρακαλώ και από τη Λισαβόνα μέχρι το Λίνεμπορχ της Γερμανίας. Γιατί μας παρακολουθεί η Ευρώπη. Φυσικά έχουμε και διερμηνία και σας παρακαλώ να μιλάτε όλοι καθαρά και αργά για να μπορούν οι μεταφράστριες και οι μεταφραστές να σας παρακολουθούν και να κάνουν τη δουλειά τους με ωραίο τρόπο. Ε, ε, ε, Μετά, στην ομάδα ENF έχουμε μια αλλαγή. Ο κύριος Λανκίνη έρχεται να αντικαταστήσει τον κύριο Σαλβίνη. Και πάμε στο σημείο 3. παρουσίαση τη καταρχή Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού και μάλιστα εξυγχρονισμό τη συμφωνία. Στις 21 Απριλίου συμφωνήθηκε επί της αρχής λίγο πριν από την έκθεση του Ανοβέρου που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου και φέτος συμμετέχει και το Μεξικό ως εταίρος ε, της έκθεσης ε, του Ανοβέρου. Οπότε ήταν και πολύ καλή η ευκαιρία αυτή. Να παρουσιαστεί καταρχήν συμφωνία και να ε, καταδείξουμε τις σχέσεις που έχουμε με το Μεξικό. Και βεβαίως ζούμε σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο με τις παλινοδίες του κύριου Τραμπ θα πρέπει να πούμε ότι εμεί θέλουμε εμπόριο με βάση κανόνες και το διατρανώνουμε με τον καλύτερο τρόπο έτσι. Έχουμε και επισκέπτες σήμερα για το σημείο αυτό και θέλω να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον πρέσβη, τον νέο πρέσβη του Μεξικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκανέρο λέγεται. Καλωσορίσατε. και τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Μεξικού, τον κύριο Γκέρα και τους επικεφαλής ε, την επικεφαλής μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Κιονίχη. Και έχουμε και μόνιμο εισηγητή για τις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό και τις εμπορικές συμφωνίες που είναι η συγκεκριά η κυρία Ροντρίγκε Πίνερ. Θα ήθελα να παρακαλέσω πρώτα την κυρία Κένιχ να μας παρουσιάσει λίγο το θέμα και τι σημαίνει αυτή η καταρχήν συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Και το χρονικό ορίζοντα. Παρακαλώ, κυρία Κένιχ. Thank you very much, Chairman, and uh, I'm very happy to be. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και πολύ χαιρόμαστε που στις 21 Απριλίου καταφέραμε να καταλήξουμε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικό. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν περίπου δύο χρόνια. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πήγαν γρήγορα διαπραγματεύσεις και ήταν ιδιαίτερα εντατικές. Καταλήξαμε λοιπόν και σίγουρα χρειάστηκε κάποια πίεση, τα καταφέραμε. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Μεξικό θέλουν να ενισχύσουν το διεθνές εμπορικό σύστημα, θέλουν καλές συμφωνίες για να αναπτυχθεί παρετέρω το εμπόριο και να δοθεί όθηση στο γενικότερο εμπορικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας τώρα. Θα είδατε ότι δημοσιεύσαμε την καταρχήν συμφωνία και ότι δημοσιεύσαμε και στην ιστοσελίδα μας το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αμέσως μετά την κατάληξη της συμφωνίας. Κάποια κομμάτια κειμένου δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Τα δουλεύουμε. Όπως θα θυμόσαστε και από άλλες τέτοιες καταρχήν συμφωνίες, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες τακτοποιούνται την τελευταία στιγμή ακριβώς γιατί οι διαπραγματεύσεις κράτησαν λιγότερο από δύο χρόνια, υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που θα έπρεπε να χτενιστούν λίγο. Οι λεπτομέρειες δηλαδή για προθεσμίες, για καταλόγους ε, γεωγραφικών ενδείξεων κτλ. Τώρα αυτά στο οποία καταλήξαμε είναι σημαντικές πολιτικές λεπτομέρειες Τίποτα δεν έχει μείνει άλυτο, το οποίο κινδυνεύει να πειράξει την ισορροπία αυτή της συμφωνίας. Τι πετύχαμε με τη συμφωνία αυτή είναι πολύ φιλόδοξη. Θα θυμόσαστε ότι είχαμε μια συμφωνία η οποία λειτουργούσε ικανοποιητικά, αλλά υπήρχαν κάποιες αδυναμίες και λήψει γιατί δεν καλύπτονταν ακριβώς όλα τα ζητήματα τα οποία κανονικά καλύπτονται από εμπορικέ συμφωνίες. Πρόσβαση στην αγορά, δεν υπήρχαν τα γεωργικά προϊόντα μέσα, ούτε τα μεταπημένα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο εξυγχρονισμού τη συμφωνία. Και ένα δεύτερο τομέα ήταν εκείνο των υπηρεσιών έχουν γίνει στο Μεξικό σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θέλαμε να συμπεριλάβουμε στη νέα συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ελευθέρωση πολλών υπηρεσιών εκεί. Και πιο συγκεκριμένα έγιναν αλλαγές στις υπηρεσίες στο θαλάσσιο χώρο, στις τηλεπικοινωνίες και αλλού, πολύ σημαντικοί τομείς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, Επίσης έχουμε και ένα κεφάλαιο όσον αφορά τις επενδύσεις και την προστασία των επενδύσεων. Εκεί έχουμε καλά αποτελέσματα γιατί το Μεξικό είναι έτοιμο να δουλέψει με ένα σύστημα μόνιμων διαιτητικών ε, επενδυτικών ε, δικαστηρίων και έχει δεσμευτεί για το σύστημα αυτό πλήρως. Ενισχύονται επίση οι κανόνε για τι επενδύσει. Συμφωνήσαμε επίση με το Μεξικό ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα πολυμερέ ε, διαιτητικό δικαστικό σύστημα όσον αφορά τις επενδύσεις. Αυτό το προετοιμάζουμε. Και πιστεύουμε ότι είναι και αυτό θετικό. Εξετάσαμε και τα μη δασμολογικά τους μη δασμολογικούς φραγμούς που υπάρχουν ανά τον κόσμο και είναι μερικές φορές πιο σημαντικό να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα γιατί δεν πρέπει η πρόσβαση στην αγορά ε, να αντιμετωπίζει άλλο είδους προσκόμματα πέρα από τους δασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και εμείς έχουμε δεσμευτεί υπέρ της ρύθμισης με την αρχή της προφύλαξης που αποτελεί στοιχείο κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι ναι, δεν θέλουμε ε, μη δασμολογικούς φραγμούς, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και εμποδίζουν τους καταναλωτές. Εξετάζουμε μη δασμολογικούς φραγμούς και στον ε, φυτογενομικό και υγειονομικό τομέα. Και εδώ ε, υπάρχουν διάφορα ζητήματα στην εφαρμογή της τρέχουσας συμφωνίας με την πλευρά του Μεξικού είχαμε πολύ καλή συνεργασία και προσπαθήσαμε να λύσουμε διάφορες δυσκολίες που είχαμε στα φυτοϊγειονομικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ε, SPS. Οπότε ε, φροντίσαμε να προχωρήσουμε και για την επόμενη συμφωνία αλλά και να εφαρμόζεται η τρέχουσα συμφωνία όσο γίνεται καλύτερα στο κομμάτι που αφορά το SPS. Η συμφωνία καθορίζει και ισότιμες συνθήκες για τα δικαιώματα διονυτικής ιδιοκτησίας. Θα έχουμε περισσότερη συνεργασία για να καταπολεμήσουμε καταχρηστικές πρακτικές και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και για τις γεωγραφικές ενδείξεις, όπου υπάρχει προστασία για τουλάχιστον 340 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις. Όπως θα θυμόσαστε και από άλλες συμφωνίες και εδώ, ήμασταν προσεκτικοί. Είχαμε μια καλή συζήτηση με το Μεξικό για ειδικέ γεωγραφικές ενδείξεις όπου υπάρχει ε, θεμητό εμπόριο με το Μεξικό, οπότε όπως κάναμε και σε άλλες συμφωνίες και εδώ καταλήξαμε σε ειδικέ λύσεις για μερικές γεωγραφικές ενδείξεις σχετικά με τις οποίες οι παραγωγοί και οι καταναλωτές στο Μεξικό είχαν ε, θεμητά συμφέροντα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεχίσουν να παράγουν. Για την πρόσβαση στην αγορά, όπως είπα και νωρίτερα, δεν είχαμε συμπεριλάβει πριν ε, ούτε τα ε, γεωργικά προϊόντα, ούτε τα μεταποιημένα. Ε, Τώρα συμπεριλαμβάνονται και αυτά. Και έχουμε κάποιες δασμολογικές ποσοστώσεις για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκές ευαισθησίες, αλλά και ευαισθησίες από την πλευρά του Μεξικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε μια καλή και ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά και για προτεραιότητας προϊόντα, όπως είναι τα πουλερικά ή το χείριο κρέας. Μια άλλη δυσκολία θα τα είδατε και στον τύπο. Το Φεβρουάριο προσπαθήσαμε να καταλήξουμε για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά υπήρχαν δυσκολίες. Για το ευρωπαϊκό εμπόριο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για το Μεξικό. Στο τέλος καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία γενικού χαρακτήρα που προστατεύει το 45% το δικό μας επίπεδο για πρώτες ύλες με κάποια ευελιξία για τους Μεξικανούς παραγωγούς για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και εμείς αξιολογούμε το αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό και, και για τις δύο πλευρές και προστατεύει σίγουρα τα ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα της ευρωπαϊκής δηλαδή αυτοκινητοβιομηχανίας για τις ε, δημόσιες προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις. Θα θυμόσαστε ότι όταν είμαστε κάτω από το ομοσπονδιακό επίπεδο ε, δεν υπήρχε κάλυψη στην προηγούμενη συμφωνία. Συζητήσαμε επί μακρό με το Μεξικό επ' αυτού. Ποτέ δεν είχε δεσμευτεί για ένα κεντρικό επίπεδο το Μεξικό. Αλλά ακριβώς ε, σε αυτό χρειάζεται απόφαση από την κεντρική αρχή. Τώρα, και δεδομένων και των εκλογών, το Μεξικό συμφώνησε και ξεκίνησε ήδη διαβουλεύσεις με τις διάφορες περιφέρειες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για πρόσβαση στις αγορές όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι ένα επίπεδο ε, του ΑΕΠ των ε, περιφερειών αυτών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, οι διαβουλεύσεις θα τελειώσουν μάλλον στις αρχές του 2019, το νωρίτερο. Όπως και να έχει το πράγμα, θα ολοκληρωθούν πριν να έχουμε τελειώσει και με το τεχνικό σκέλος, τη μετάφραση, έτσι ώστε να παρουσιαστεί συμφωνία στις χώρες μέλη και στο Κοινοβούλιο που είναι πολύ σημαντικό για μας. Και θα είμαστε σε επαφή με το Μεξικό σε όλη τη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ας κοιτάξουμε λίγο τώρα το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση με το εμπόριο. Εδώ, ως ήθιστε υπάρχει το δικαίωμα στην ρύθμιση, υπάρχει αρχή της προφύλαξης, όπως είπα και πριν, που ισχύουν και εδώ, και έχουμε δέσμευση απέναντι και στις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και πρέπει να υπάρξει και κύρωση των ε, συμβάσεων όπως είναι 98 που δεν έχει ακόμα κυρώσει το Μεξικό. Ε, κρεμεί πρόταση στη Γερουσία εδώ και αρκετό καιρό και εμείς θα παρακολουθήσουμε και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις όσον αφορά την κύρωση και τη σύμβαση αυτής. Επίσης, έχουμε δεσμευτεί για την εφαρμογή περιβαλλοντικών συμφωνιών για το εμπόριο και την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένης και τη Συμφωνία των Παρισίων, βιώσιμη ε, ανάπτυξη και αλυσίδες προμήθειας, προστασία του θαλάσσιου χώρου και καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριας πανίδας. Ως ήθιστε επίσης, η εφαρμογή κεφαλαίων θα περάσει από διαβούλευση αλλά και από πάνελ εμπειρογνωμόνων και θα γίνουν και παρουσιάσεις εκθέσεων. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θέλω επίσης να αναφέρω ότι στη συμφωνία αυτή που είναι σύνδεσης, έτσι, υπάρχει το πολιτικό σκέλος η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα θα εξετάσει το σύνολο της συμφωνίας ε, σύνδεσης, όλα τα κεφάλαια δηλαδή. Θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ε, θέματα από το σύνολο της συμφωνίας σύνδεσης, κάτι το οποίο είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και έχουμε και ένα μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών και από τις δύο πλευρές. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει παράρτημα για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις διάφορες αρχές, τις διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες είναι συμβαλόμενα μέρη τόσο το Μεξικό όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στα πλαίσια του ΟΗΕ, αλλά και σε σχέση με τους στόχους του 2030 για τους βιώσιμους στόχους. Η υλοποίηση του παραρτήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς περνάει από διαβουλεύσεις και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα και από πλευράς του Μεξικού. Τέλος, πώς προχωράμε. Όπως είπα και στην αρχή, το αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε καταλήξει της καταρχήν συμφωνίας καλύπτει όλα τα σημαντικά. Παραμένουν κάποιες λεπτομέρειες. Οι συζητήσεις για τις λεπτομέρειες θα μας πάρουν κάποιες εβδομάδες ακόμα. Και μετά θα περάσουμε στην νομική εξέταση, στο νομικό χτένισμα, που Ελπίζουμε να πάει γρήγορα. Συνήθως χρειάζονται κάποιοι μήνες, αλλά εξαρτάται βέβαια ε, οι δύο πλευρές πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν και θα συμφωνήσουν. Μετά η συμφωνία θα πρέπει να μεταφραστεί, κάτι το οποίο και αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Συνεπώς, για το χρονοδιάγραμμα, θα προσπαθήσουμε οι τεχνικές συζητήσεις, αναθεωρήσεις να ολοκληρωθούν σε δύο μήνες περίπου και μετά θα πάμε στο νομικό χτένισμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί φέτος. Αλλά πάντα υπάρχει ερωτηματικό. Έτσι εξαρτάται πόσο δύσκολο θα αποβεί το χείρημα αυτό. Η μετάφραση, απ' την άλλη, χρειάζεται 5-6 μήνες, καμιά φορά και λίγο παραπάνω. Που σημαίνει ότι θα παρουσιάσουμε την τελική συμφωνία γύρω στο 2019 Στις χώρες μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εννοείται ότι εργαζόμαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ωραία, αυτά. Και από εκεί και πέρα, αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κερνίκ. Μια συμπληρωματική ερώτηση πρώτα. Σκοπεύετε να παρουσιάσετε το εμπόριο ε, σε αγαθά και υπηρεσίες και τις επενδύσεις ταυτόχρονα ή έχετε προβλέψει διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικές ταχύτητες για να επιταχυνθεί το ένα σκέλος, το γενικό δηλαδή, και το άλλο να έρθει λίγο αργότερα για τις επενδύσεις. Thank you. That, that's a very good... Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ερώτηση. Μια που πρόκειται για συμφωνία σύνδεσης, το σύνολο της συμφωνίας θα παρουσιαστεί ως ένα, τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς. Ο μόνιμος εισηγητής μας τώρα, η κυρία μάλλον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ τον πρέσβη του Μεξικού και την ομάδα του και την κυρία Κόνη και την ομάδα της εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η συμφωνία, αυτή η καταρχήν συμφωνία έρχεται την καλύτερη δυνατή στιγμή. Διότι με αυτή τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό στέλνει ένα σαφές ε, μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ κάποιοι είναι υπέρ του προστατευτισμού και ε, να ξεκινήσουν ε, ε, φυρικτούς ε, εμπορικούς πολέμους που όλοι ξέρουμε πώς αρχίζουν αλλά ποτέ πώς τελειώνουν, αυτή η συμφωνία υποδηλώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού για ένα καθολικό εμπόριο, δίκαιο εμπόριο, το οποίο βασίζεται σε κανόνες. Και έτσι εξυγχρονίζουμε και τις εμπορικές μας σχέσεις με το Μεξικό, οι οποίες είχαν κατακαιρματιστεί από την παρούσα συμφωνία του 1999, διότι πολλά πράγματα άλλαξαν έκτοτε και επιμε... Ε, ε, ενισχύουμε τους δεσμούς μας με την Λατινική Αμερική και ε, σε διεθνές επίπεδο. Και θα ήθελα να σταθώ σε ένα στοιχείο το οποίο δεν παρουσιάζεται πολύ συχνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική από κοινού είναι το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% του ε, εσωτερικού ε, εγχώριου προϊόντος. Και το Μεξικό είναι η δεύτερη χώρα στη Λατινική Αμερική σε οικονομικά στοιχεία και σε πληθυσμό. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, διευρύνουμε, να εμβαθύνουμε τις οικονομικές πολιτικές μας και εμπορικές μας σχέσεις και να τις χρησιμοποιήσουμε στα διεθνή βήματα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε αυτή την πιο δίκαιη ε, συνεργασία στην οποία προσβλέπουμε όλοι. Και θα ήθελα να σταθώ και στις προσπάθειες που έκανε το Μεξικό για να απαντήσει σε κάποια περίπλοκα ζητήματα, ε, ξεκινώντας μάλιστα και από τελείως διαφορετικές ε, θέσεις από αυτές στις οποίες καταλήξαμε τελικώς. Αναφέρομαι στη νέα πολιτική επενδύσεων, την οποία υπερασπιστήκαμε εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν ήταν η αρχική θέση του Μεξικού όσον αφορά το σύστημα τη διαιτησία. και αναφέρουμε επίση και στην αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων. Πιστεύω ότι η στάση του Μεξικού ήταν ε, ε θετική και θα ήθελα για άλλη μια φορά να το επισημάνω και επίσης οι προσπάθειες που έκαναν όλες οι πλευρές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πράγματι ε, δύο χρόνια είναι χρόνος ρεκόρ για την επίτευξη ε, του εξυγχρονισμού μιας συμφωνίας τόσο ευρείας όσο αυτή. Και θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημαντικά επιτεύγματα. Καταρχά, ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται σε εμπορική συμφωνία ένα κεφάλαιο καταπολέμηση τη διαφθοράς. Θεωρώ ότι αυτό είναι πρωταρχική σημασίας και είναι και πρωταρχική σημασίας διότι θέλουμε να βοηθήσουμε το Μεξικό να πετύχει ε, να καταπολεμήσει ε, τη διαφθορά, αυτή τη μάστιγα την οποία πληρώνουν οι Μεξικανοί αλλά και όλοι. Επίσης ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε από κοινού τη διαφθορά όπως είπα αλλά και το ξέπλυμα χρήματος και σε εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο η προστασία 340 γεωγραφικών ενδείξεων ε, της Ευρώπης οι οποίες ε, ε, κυριαρχούν στη μεξικανική αγορά είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα όπως επίσης και η πρόσβαση στην αγορά δημοσίων προμηθειών στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Κόνιγκ και η οποία είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δέσμευση για το άνοιγμα των αγορών σε υποπεριφερειακό επίπεδο κατά την υπογραφή της συμφωνίας που θεωρώ ότι είναι στρατηγική σημασία. Επίσης μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο είναι καινοτομία. Και για πρώτη φορά θα έχουμε μια εμπορική συμφωνία με ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολλά τα επιχειρήματα τα οποία ακούμε ε, και ε, είναι και κενά νοήματος ε, από μια μεριά. Ε, οι εμπορικές συμφωνίες λέγεται πάντα ότι ευνοούν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί οι μεγάλες πολυεθνικές δεν χρειάζονται εμπορική συμφωνία. Εγκαθίστανται απευθεία εκεί που τους βολεύει περισσότερο και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν όλα τα διοικητικά προβλήματα και όλα τα θεσμολογικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από το εμπόριο. Το γεγονό λοιπόν ότι εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι αυτές οι οποίες αποφελούνται περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία και ότι υπάρχουν όλα τα μέσα προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την εμπορική αυτή συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι οι εμπορικές συμφωνίες ε, δεν είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύονται οι κυβερνήσεις. Το διαπραγματεύονται οι κυβερνήσεις για να ευνοήσουν τον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ενισχυμένος διάλογος και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί καινοτομία από το σύνολο των διατάξεων της συμφωνίας. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί ένα τεράστιο άλμα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει και υπόδειγμα για όλους τους υπολείπους διότι δεν είναι μόνο το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης όπως ε, γίνεται συνήθως Αυτά λοιπόν είναι τα επιτέχματα τα οποία ήθελα να επισημάνω ως πιο σημαντικά και είναι και τα θέματα τα οποία ανέκαθεν αποσχολούσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ε, λογικά φυσικά υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες ε, μεταξύ των οποίων θα ήθελα να ε, τονίσω τα εξή. όσον αφορά το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης. θα υπάρχει ίδιος ε, σεβασμός για τα κοινωνικά, εργατικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα όπως ε, υπάρχει και στη συμφωνία με τον Καναδά. Το Μεξικό, όπως πολύ σωστά επεσήμανε η κυρία Κόνιγκ, ακόμα δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση 98 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ε, δεν έχει σημασία μόνο ε, να υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες και να υπάρχει εμπόριο, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία, διότι το εμπόριο αποτελεί μέσο για την ανάπτυξη, μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσο ε, για τη δημιουργία ευημερίας, Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, υπό ποιε κοινωνικέ, εργατικέ και περιβαλλοντικέ συνθήκε ε, γίνεται όλο αυτό. Και φυσικά μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική η δέσμευση από πλευρά των Μεξικανικών Αρχών για την κύρωση τη Σύμβαση 98 και την εφαρμογή της ε, σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, είπα ότι είναι θετικό το γεγονός ότι γίνεται μια αλλαγή για το Μεξικό που είχε ένα σύστημα το οποίο δεν βασίζεται σε γεωγραφικές ενδείξεις αλλά στο εμπορικό σήμα και το γεγονός ότι αναγνωρίζει το κατάλογος ε, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες διότι κάποιες από τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα μπορούσα να σας αναφέρω ε, το Μαντσέγκο, αλλά υπάρχουν και άλλες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ιταλία και από την ε, Γαλλία. Βάσει του συστήματος λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση ότι δεν θα γίνει κανένα ε, σφάλμα για τον καταναλωτή όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος. Υπάρχει για παράδειγμα παραγωγή του Μαντσέγκο και στο Μεξικό. Αλλά δεν είναι το ίδιο προϊόν με αυτό το οποίο παράγεται στην Καστίγια Λαμάντσα στην Ισπανία και φυσικά η προστασία ε, σημαίνει ότι στην ετικέτα θα ε, γίνεται διάκριση σαφή μεταξύ των προϊόντων, θα λέγεται ότι είναι τελείω διαφορετικά προϊόντα για να μην παραπλανά το καταναλωτέ. Και το θέμα είναι πώς θα ελεγχθεί αυτό στην πράξη, ότι όντως τηρούνται οι δεσμεύσει τη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Η κυρία Κόνικ είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά ε, στοιχεία περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά στο ε, φύλλο. Ε, είναι όντως αυτό ε, το να συμπεριλαμβάνουμε τα πολιτικά στοιχεία. Καμία συμφωνία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να παραβλέπει το μισό πληθυσμό ε, του κόσμου και θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στις ε, διατάξεις όσον αφορά το φύλλο. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται αυτό, αλλά με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Συμφωνία Σύνδεσης δεν είναι δημόσια. Έχει δημοσιοποιηθεί όντως, υπάρχουν στο διαδίκτυο τα κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνονται, αλλά δεν είναι έτσι μια συμφωνία σύνδεση. Κάνω έκκληση προς όλους να υπάρχει διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Thanks a lot uh, for this first... Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη αυτή ε, εκτίμηση ε, της διαδικασίας. Σκιώδης τώρα. συγητές ε, Και μετά έχουν ζητήσει κάποιοι βουλευτές το λόγο. Ε, να βάλουμε και ένα όριο, δύο λεπτά. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κανονικά είναι ο κύριος Φίσας. Τον αντικαθιστά κανείς, όχι. Η κυρία Μακλάκλιν, επίσης απούσα. Ε, η Τίτα Σαράνσοβα από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσμα. Ε, τώρα καταφέραμε πραγματικά να εξυγχρονίσουμε τη συμφωνία που έχουμε με το Μεξικό. και εμείς είμαστε εκείνοι που υποστηρίζουμε την ε, περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου. Υπάρχει ένα θέμα που με ανησυχεί λίγο. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η συμφωνία. Είναι κρίμα αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε μια συμφωνία, να μην λαμβάνουμε υπόψη όλα τα σημαντικά στοιχεία και εννοώ σημαντικά για τις επιχειρήσεις των 21ο αιώνα δεν υπάρχουν ουσιαστικές ε, ε, πρόνοιες για την ε, ροή δεδομένων και πληροφοριών με το Μεξικό. Είναι κρίμα. Έχουμε αντίστοιχη εμπειρία με την Ιαπωνία. Γιατί δεν καταφέραμε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο φιλόδοξο στη συμφωνία με το Μεξικό. Θα ήθελα να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το χρονοδιάγραμμα, μήπως θα μπορούσατε να είστε πιο συγκεκριμένοι. Πώς βλέπετε τώρα την πορεία από εδώ και πέρα. Μιλήσατε για τη μετάφραση. Ωραία. Με πραγματικούς όρους πότε πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Χάιντι Χάουταλα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Βεβαίως έχει έρθει η ώρα του εξυγχρονισμού ε, της συμφωνίας με το Μεξικό, αλλά η δική μου ομάδα εξεκολουθεί να έχει πολλές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, πώς δένουμε τα χέρια των επόμενων κυβερνήσεων με αυτή την καταρχήν συμφωνία ε, τη επόμενη συγκεκριμένα κυβέρνηση, γιατί η συμφωνία γίνεται ε, μεσού τη προεκλογική εκστρατεία και 1η Ιουλίου έχουν εκλογές. Τι περιθώριο ε, χειρισμών θα έχει η ιουλιου εχουν εκλογέ. τι περιθωριο χειρισμων κυβέρνηση με την καταρχήν αυτή συμφωνία. Ένα αυτό δεύτερο. Αν καταλαβαίνω σωστά το κείμενο, στο άρθρο 22 παράγραφος 4 στην καταρχήν συμφωνία ορίζεται ότι ένας επενδυτής μπορεί να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη συμφωνία και να ζητήσει αποζημίωση αν βλάπτεται, ε, ακόμα και αν δεν έρθει ποτέ η οριστική συμφωνία. Αυτό πώς εξηγείται. Στη συνέχεια, μας εξηγήσετε πάρα πολύ λεπτομερώς ε, το ε, περιεχόμενο του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά δεν μένει ικανοποιεί πάρα πολύ αυτά αυτό που ακούω για καταλόγους και ε, τις διεθνείς και τη σύμβαση του 96, το ΑΕΛΟ που ακόμα δεν έχει ε, κυρωθεί ε, και αφορά τη ε, διαφάνεια και την χνηλασιμότητα ε, στην διατροφική αλεξίδα. Και ωραία είναι αυτά που λέτε για τη βιωσιμότητα και για την βιοπικιλότητα, αλλά το να παριθμούμε κάποιους καταλόγους συμβάσεων και νομοθεσία σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν κιόλα. Και τέλος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλήματος χρήματος. Υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες καταγγελίες, για παράδειγμα της τράπεζας Rabobank για ξέπλυμα χρήματος. Τι θα κάνετε με το τελικό κεφάλαιο για την καταπολέμηση αυτών από την ε, Ενωτική Αριστερά. Η Λόλα κανονικά, αλλά η κυρία Μινόερ τώρα. Παρακαλώ. Στα αγγλικά. Α, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχώς επαναλαμβάνει και τώρα εδώ ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι ε, ε, Αυτό ελέγχεται. Ε, τι, τι γίνεται με το κλάδο της ε, ε ενέργειας. Λένε ε, οι δημοσκοπήσεις ότι θα ε, ιδιωτικοποιηθεί η ενέργεια και θα υποφεληθούν και τρέχουν να υποφεληθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Ποια είναι τα αμοιβαία ωφέλη. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας λέει ε, θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ως προς τη βιωσιμότητα πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτό δεν έχει γίνει. Πώς υπογράφεται η συμφωνία καταρχήν. Θέλω να παρακαλέσω την εισηγήτρια να ασκήσει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια, η διαφθορά είναι μεγάλο πρόβλημα ε, και ε, η εγκληματικότητα σχετικά με τα ναρκωτικά. Γιατί δεν έχετε εφαρμόσει ποτέ τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και το νέο κεφάλαιο για την καταπολέμηση της διαφοράς, πώς θα επιβληθεί, υπάρχει μηχανισμός επιβολής κυρώσεων αποτελεσματικός δεν έχουν κυρώσει επίση τη σύμβαση του Διεθνού Οργανισμού εργασία ε, ε, το 1996 και πώ θα του υποχρεώσουμε να το κάνουν. Και τέλο είπατε ότι α, υπάρχουν και κάποιε λεπτομέρειε που πρέπει να διεκπαιρεθούν. Ξέρουμε όμω ότι ο διάβολο εκεί κρύβεται στι λεπτομέρειε. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πότε θα τα συζητήσετε και γιατί δεν τα έχετε ακόμα διεκπαιρεώσει αυτά τα θέματα που τα λέτε στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ εγώ. Η Καρολίν Grandfather Heinz. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, χαίρομαι και εγώ. Το βρίσκω πολύ θετικό για τη ρήτρα κατά πολέμηση διαφθορά. Και ποια εργαλεία χρειάζομαστε για να μπορούμε να το επιβάλλουμε κιόλα γιατί νομίζω είναι μια διαδικασία διαβούλευση αυτή που προβλέπετε. Μετά η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ θετικό επίση και στη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά δεν ξέρουμε και πάλι πώ θα έχει διαδικασία. Αν κάποιο, α πούμε, θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, πού θα αποτανθεί και ποιο αποφασίζει για το παραδεκτό και για την αναστολή των ε, εμπορικών προτιμήσεων και συμμετέχει αυτό στη διαδικασία επίλυσης διαφοράς. Δεν υπάρχουν εργασιακά πρότυπα, είπαμε δεν έχουν κυρωθεί όλες οι συμβάσεις ILO. Όταν θα υπογραφεί η συμφωνία, θα έχουν κυρωθεί όλες αυτές οι συμβάσεις και αν δεν κυρωθούν δεν θα τα υπογράψουμε και το κεφάλαιο για την βιωσιμότητα. Για μένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι μηχανισμοί κυρώσει. Ξέρουμε τι παθαίνουν εκεί οι δημοσιογράφοι, τα συνδικάτα και οι ΜΚΟ που διώκονται έως και θανατώνονται. Τι θα γίνει λοιπόν αν δεν έχουμε μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων και ε, την προστασία του περιβάλλοντος. Θυμάμαι ακόμα ε, ένα πρώην συνάδελφο το Σόριν Νόισερ που ήταν και αρμόδιος για αυτό το θέμα, που επέμενε πάρα πολύ να υπάρξει μηχανισμός κυρώσεων, αλλά αυτό δυστυχώς χάθηκε. Και ποιος θα προστατεύει τα δικαιώματα. Και η αρχή της προφύλαξης στο κεφάλαιο της αηφορίας και της βεσιμότητας δεν αναγράφεται πουθενά. Όταν έχουμε λοιπόν παραβιάσεις και παραβάσεις, πώς θα τις διαπιστώνουμε και πώς θα επιβάλλουμε κυρώσεις. Ευχαριστώ και τηρήστε απολύτως και το χρόνο σας. Η Μαρία Γενά. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Την ίδια ερώτηση έχω και εγώ για τις εκλογές της 1ης Ιουλίου. Τι περιθώριο λιγμών υπάρχει άπαξ και αλλάξει η εξουσία ε, σε σχέση με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις της συμφωνίας αυτής. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών ε, αν έχουμε νέα πολιτική εκπροσώπηση που έχει εκλεγεί και που δεν έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το περιθώριο. Δεύτερον, αν ε, δούμε την ε, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό, διαπιστώνουμε ότι υπήρχε ρήτρα για το δικαίωμα στην εργασία, για, το, για την εργασία των παιδιών και για την ασφάλεια στην εργασία οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν επειδή οι επιχειρήσεις δεν σέβονταν αυτές τις παράλληλες συμφωνίες και δυστυχώς ποτέ δεν κατέληξαν αυτές οι διαμαρτυρίες γιατί η συμφωνία δεν προέβλεπε μηχανισμό κυρώσεων αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο. Εσείς το έχετε σκεφτεί, έχετε προβλέψει κάτι για αυτή τη συμφωνία. Τρίτον, το μείγμα της συμφωνία. Ξέρω ότι 22 Μαΐου γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο για τη νέα δομή των εμπορικών συμφωνιών. Για τη συμφωνία αυτή θα συνεχίσετε να δουλεύετε στα πλαίσια ενός μοντέλου μικτού ή θα προτείνετε διαχωρισμό των διατάξεων. Για το ICS, εσείς ε, συνεχίσετε να δουλεύετε όπως και με τη συμφωνία με τον Καναδά, ενώ εκεί για τον Καναδά δεσμευτήκατε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσετε όσα υπάρχουν στη συμφωνία με τον Καναδά. Τι γίνεται τώρα με αυτή τη δέσμευση που πήρατε και για την βιώσιμη ανάπτυξη προτείνεται να έχετε ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ εδώ έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, καμία βελτίωση. Είσαστε στο status quo. Ευχαριστούμε. Κύριε Σούστερ, ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί με κάλυψαν οι ερωτήσει. Δύο είναι τα ουσιαστικά ερωτήματα. Είναι προπόθεση ε, η συμβάσεις στο ILO να εγκριθούν και να κυρωθούν πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ή γίνεται απλώς μια ασαφής αναφορά ότι στο μέλλον πρέπει να το κάνετε. Γιατί με τέτοιε δηλώσει προθέσεων έχουμε κακές εμπειρίες στο παρελθόν. Και το δεύτερο, με τη δυνατότητα επιβολής και εφαρμογή, είχαμε μακρά συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητα επιβολής ε, κεφαλαίων βιωσιμότητας σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες. Και τι έχει βελτιωθεί τώρα στη συμφωνία με το Μεξικό σε σχέση με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες. Πολύ σημαντική ερώτηση. Ο κύριος Ρεμπίχη. Ευχαριστώ. Μία από τις ερωτήσεις είναι ακριβώς πώς ε, υπολογίζονται οι ροές των αγαθών. Έχουμε στη Σεβίλη ένα κοινό κέντρο ερευνών ε, που ε, τα μετράει αυτά. Στη συμφωνία με τη Νότια Κορέα μάθαμε ότι το κέρδος ε, ήταν ε, στην ε, αύξηση της κυκλοφορίας των αγαθών 30% και παραπάνω και για τις δύο πλευρές. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δημιούργησε και θέσεις εργασίας και βημερία. Εδώ το υπολογίζουμε πώς θα μεταφραστεί αυτό σε θέσεις εργασίας. Για την επιβολή όλων αυτών των διατάξεων και των κυρώσεων εξαρτώμαστε πάρα πολύ από την δικαιοσύνη τη μεξικανική. Βέβαια, εμεί εμπιστευόμαστε τα μεξικανικά δικαστήρια, αλλά ακούτε και μια δυσφορία γενικότερα. Και σε περίπτωση που δεν τα καταφέρνει η μεξικανική δικαιοσύνη, ε, τι πιστεύετε για τα διαιτητικά δικαστήρια που ορισμένοι εδώ πέρα τα απορρίπτουν. Και τελευταία ομιλήτρια η κυρία Ζαμι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη κι εγώ. Είναι προφανές ότι κυρία Συγγέντρια το μήνυμα που δίνεται στον υπόλοιπο κόσμο για μας είναι προς το κλάδο του βόηου κρέατος. Με τρόπο που καταστρέφεται ο κλάδος αυτός. Οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλους. Οι αυξητικές ορμόνες ε, στις ζωοτροφές ή προϊόντα τα οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη που χρησιμοποιούνται όμως στο Μεξικό. Αυτό δημιουργεί βέβαια ένα προβληματισμό για την υγεία, για, την υγεία, για τα φυτογειονομικά και για την αρχή της προφύλαξης. Οπότε, πώς θα γίνεται η γνηλασιμότητα στις ετικέτες. Και αναφερθήκατε και στην διαφθορά. Ωραία. Οι ετικέτες τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να αναγράφονται λεπτομέρειες στι ετικέτες στα προϊόντα που προέρχονται από το Μεξικό. Οι ετικέτες αυτές όμως περνάνε από μια διαδικασία αρνητική γιατί υπάρχει νομολογία με τις ΗΠΑ ε, ήδη και πάντα χάναμε ε, βάσει της αρχής της μη διάκρισης. Ε, ανάλογα με το τι λέει η ετικέτα για το που έχει εκτραφεί το ζώο, που έχει σφαχτεί κτλ. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής. Όμως ε, το σύστημα που χρησιμοποιεί η Γαλλία πρέπει να εξεταστεί σε αυτή την περίπτωση για να δούμε όταν υπάρχουν διαφωνίες να μην υπάρχει αυτή η αρχή της μη διάκρισης που υπερέχει αλλά η αρχή της προφύλαξης. Να λοιπόν ένα βασικό στοιχείο για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, να μας διευκρινίσετε, να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι σας. Γιατί όπως το έλεγε και η συγκεκριά μας, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να γίνεται θύμα κοροϊδίας. Θα πρέπει να ξέρει, γιατί στο κάτω-κάτω ε, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι επιλογές του. Είτε είναι για λόγους υγείας, είτε όχι. Ωραία. Ο νέος πρέσβης, ο κύριος Σασκανέρο τώρα, παρακαλώ, να πάρει το λόγο. Το πολύ πέντε λεπτά όμως παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ και σας και τα μέλη της Επιτροπής αυτής για την ευκαιρία που ε, μου δίνετε να έρθω εδώ να ακούσω τις συζητήσεις σας και να απευθυνθώ σε σας. Ως νέος πρέσβης του Μεξικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρία που είναι η πρώτη συνεδρία τη Επιτροπής σα μετά την κατάληξη της καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού. Για μα αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση στρατηγική σημασίας και οικονομική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. Η συμφωνία, όπως γνωρίζετε, είναι μια συμφωνία συνολικής κάλυψης. Μια φιλόδοξη και καινοτόμα συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Πρώτον, ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου. Διάρθρωση του πολιτικού διαλόγου στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μας με την βοήθεια των ε, βουλευτών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της. Διμερός, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού, αλλά και για να προχωρήσουμε σε κοινέ δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, η ειρήνη, ασφάλεια και η ισότιμη και διώσιμη ε, ανάπτυξη για όλους. Η συμφωνία αυτή προσφέρει λοιπόν μια βάση για ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που θα βοηθήσει το το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα με συνεργασία ε, σε τεχνικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και ε, περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να ενισχυθούν οι οικονομικοί μας ε, πόροι, ηλικοί και του ανθρώπινου δυναμικού. Στον οικονομικό τομέα, δίχως άλλο, η συμφωνία αυτή ανοίγει νέες μεγάλες ευκαιρίες για πρόσβαση στις αγορές για την διευκόλυνση των επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και θα υποφεληθούν κύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η συμφωνία λοιπόν είναι μια συμφωνία από την οποία όλοι έχουν κερδίσουν. Είναι μια συμφωνία αμοιβαία αποφελής η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη και δύο πλευρές, να διαφοροποιήσουμε τις σχέσεις μας με τον έξω κόσμο και θα μας επιτρέψει επίσης να διαρθρώσουμε καλύτερα ε, το κοινό έργο ε, Μεξικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Πάνω απ' όλα όμως η συμφωνία αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για την σημασία που έχει το ελεύθερο εμπόριο εμπόριο το οποίο να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους κοινωνικούς στόχους. Είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα επίσης υπέρ της πολυμερούς διάστασης και τον καθορισμό κοινών κανόνων, του οποίους όλοι να σέβονται. Είναι ένα μήνυμα προς την διεθνή κοινότητα ε, για το ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωριζόμαστε ως εταίροι μεταξύ μας για να οικοδομήσουμε μια νέα διεθνή διακυβέρνηση η οποία θα στηρίζει την ε, βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο για ένα κόσμο πιο δίκαιο, ε, χωρίς αποκλεισμούς, ένα κόσμο που θα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά από κοινού τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ενός κόσμου που αλλάζει όλο και περισσότερο και είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένος. Εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να σας πω ότι η πρεσβεία του Μεξικού είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να συνεργαστεί με τη σημαντική αυτή επιτροπή σας διεθνούς εμπορίου για να συσφίξουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Μεξικού και ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την, ε, τις εργασίες της αποστολής εργασίας που θα πάει αρχές Ιουνίου στο Μεξικό με την εισηγήτρια της ε, συμφωνίας αυτής την Μπακουλάδα Ροντρίγες Πινέρο, που θα συνοδεύεται και από τον κύριο Σαντιάγο Φίσας που είναι ο σκιώδης εισηγητής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν σας περιμένουμε και ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή για να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας. Πρόεδρε, θα ήθελα να επιτρέψω στον εμπορικό επιτετραμένο της πρεσβεία μας, τον κύριο Αγκέρα, να πάρει τον λόγο, που είναι υπεύθυνο για τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για το εμπορικό σκέλος της νέας αυτής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τότε Είναι πάρα πολύ σημαντική η χρονική συγκυρία στην οποία έρχεται η συμφωνία, όχι μόνο λόγω του παγκόσμιου εμπορικού πλαισίου, αλλά γιατί σπάει ο μύθος ότι ε, το Μεξικό θα έπρεπε πρώτα να συνάψει συμφωνία με τους εταίρους της ναύτας στην Αμερική και μετά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα και πιστεύουμε σίγουρα ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει αυτό. Έχουν λυθεί σημαντικά θέματα πρόσβαση ε, σε αγαθά υπηρεσίε, δημόσιε προμήθειες και νέα θέματα έχουν ενταχθεί και έχουν ληφθεί υπόψη ευαισθησίες ε, με ε, ισορροπία, όπως είπε και η κυρία Ροδρίγη Πινιέρο. Στην περίπτωση του Μεξικού, Χρειαστήκαμε ιδιαίτερες προσπάθειες να καταλάβουμε από πλευράς Μεξικού σε θέματα καινοτόμα, όπου κατανοήσαμε ότι έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει αποτελέσματα από την ε, διαπραγμάτευση αυτή. Παρόλο που είναι χορτογράφητα τα νερά αυτά, ε, συμφωνήσαμε ε, για ένα δικαστήριο διμερές για να επιλύει τις διαφορές με διαιτητικό τρόπο τύπου ΣΕΤΑ και θέλουμε ε, να πάρουμε και την εμπιστοσύνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες ε, προμήθειες στο παρελθόν, το Μεξικό είχε υποχρεώσεις μόνο σε επίπεδο επικράτειας ομοσπονδιακής. Σύμφωνα όμως και με την ΑΦΤΑ, συμμετέχουν και κάποιες από τις 32 πολιτείες τώρα σε αυτή την προσπάθεια. Κάτι άλλο που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι οι γεωγραφικές ενδείξει. Ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και ένα μικρό προηγούμενο, γιατί και οι δύο πλευρέ έχουν ένα εργαλείο το οποίο ε, προστατεύει τα ε, πνευματόδη και αλκοολούχα ποτά. Υπάρχει και μια, ένα πρότυπο ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις. 340 ε, ονομασίες ε, προέλευσης χωρίς τα ε, αλκοολούχα ποτά που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα δεν έχει εξαιρεθεί. 20 προϊόντα είναι από το Μεξικό και 19 είδη χειροτεχνίας ή παραδοσιακά στο μέλλον καλύπτονται τα γεωργικά προϊόντα, εδραιώνονται η διαρθωτική μεταρρύθμιση στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στο Μεξικό μεταξύ άλλων. Ε, εισάγουμε θέματα νέας τεχνολογίας, ε, αηφόρος ανάπτυξη, κρατικές ενισχύσεις, κρατικές επιχειρήσεις, ενέργεια, καταπολέμηση διαφθοράς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά ευημερία των ζώων είναι μερικά από αυτά. Τέλος, συμφωνώ με τον πρέσβη Εσκανέρο και είμαι στη διάθεσή σας και εγώ σε περίπτωση που έχετε περιέργεια για να μάθετε τι πιστεύει το Μεξικό ή για να διασκεδάσουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ή ανησυχία για τα εμπορικά θέματα. Δεν θέλω να μην εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εξάρω την ε, ε, θαυμάσια και αγαστή συνεργασία των δύο διαπραγματευτικών ομάδων. Ήταν πάρα πολύ σημαντική και θέλω ε, ιδιαίτερα να τονίσω την ηγετική στάση της συναδέλφου διαπραγματεύσεως κυρία Ελένα Κένικ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευγενική σας προσφορά να μας υποστηρίξετε και στο μέλλον. Είναι πολλές ερωτήσεις και τα σχόλια. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κένιχ, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Πόνσα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σύντομα για την πολιτική διάσταση του παιχνιδιού αυτού. Γιατί έχουμε και κάποια θεματάκια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάποια άλλα έτσι, πολιτικής φύσης. Sí, eh, ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί νομίζω τα περισσότερα ακούστηκαν ήδη αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος ε, σε όλους τους τομείς αυτής της συμφωνίας, που όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πρόκειται για μια καθολική συμφωνία και έχει τέσσερα κεφάλαια με ε, πολιτικά θέματα, θέματα εμπορίου και υπήρξε πρόοδο σε όλα αυτά και χαίρομαι που το διαπιστώνω. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα το πολιτικό σκέλος και το σκέλος της συνεργασίας, η νέα συμφωνία οδήγησε σε συμφωνία ήδη από το Νοέμβριο και είμαι και εγώ ικανοποιημένος, ε, διότι διαπιστώνω ότι υπάρχει συμφωνία και στο σκέλος του εμπορίου ε, που επετεύχθη στις 21 Απριλίου και όπως είπαν οι συνάδελφοι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ε, Εκκρεμούν βέβαια κάποια τεχνικά θέματα και φυσικά οι εργασίες μας συνεχίζονται σε θεσμικά και στα τελικά ζητήματα, αλλά πιστεύουμε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι θα υπάρξει συμφωνία, ιδίως σε θέματα που εκκρεμούν ακόμα στις επόμενες εβδομάδες. Και όλα αυτά φυσικά γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Και φυσικά αυτό ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο επόμενο διάστημα. Θα σταματήσω εδώ. Αν μου επιτρέπετε, αν υπάρξει οποιαδήποτε ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κόνιχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλα τα μέλη για τις πολύ καλές και πολλές ερωτήσεις. Θα δω πόσο ε, σύντομα μπορώ να απαντήσω. Να ξεκινήσω με το θέμα του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, πράγματι, οι δεσμεύσεις ε, στο κεφάλαιο του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι και αναρτημένες στο διαδίκτυο, όσον αφορά την κοινωνική εργασία, ομοιάζουν πολύ με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, αλλά υπάρχει μία διάταξη στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού, συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, για παράδειγμα, η συμμετοχή του Μηχανισμού της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία θα πρέπει να διέπει όλη τη συμφωνία. Επίσης, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά τον αντίκτυπο του εμπορίου στη βιοπικιλότητα. Υπάρχει ένα ολόκληρο άρθρο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρόκειται λοιπόν για στοιχεία τα οποία πράγματι έχουν ενισχυθεί στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού, αν τη συγκρίνουμε με τη ΣΕΤΑ. Όσον αφορά το μηχανισμό εφαρμογής, και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε πολλές συνεδριάσεις και με τους επιτρόπους. Και όπως είπα προηγουμένως, Υπάρχει ο παραδοσιακό μηχανισμός, ο οποίο υπάρχει και στις άλλες εμπορικέ συμφωνίε, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασία και βασίζεται στη συνεργασία, αλλά έχουμε και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων. Υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης ενός πάνελ εμπειρογνωμόνων επίσης και υπάρχουν και εκθέσεις οι οποίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα πεπισμένη ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος ε, να προχωρήσουμε τις ε, ε, δεσμεύσεις και να υπάρξει εφαρμογή τους και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε κυρώσεις. Δεν έχουμε δει αποτελέσματα σε συστήματα που βασίζονται σε κυρώσεις σε άλλες συμφωνίες και ακόμα και σε αυτές που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξουμε ότι μπορεί κάτι το οποίο μπορεί από το εμπόριο να έχει αντίκτυπο ε, σε συμφωνίες όπως ε, οι συμφωνίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ή κάποιες άλλες δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στη συμφωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά προβλήματα ενός συστήματος που βασίζεται σε κυρώσεις. Και φυσικά, κατά την άποψή μας, είναι πολύ πιθανότερο να υπάρχουν θετικές εξελίσεις όταν υπάρχει ε, μια ε, προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία. Και ακόμα και αν υπάρχει μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, το γεγονό ότι ε, μπορεί να δημοσιοποιηθούν εκθέσει και μπορεί να γίνει ανοιχτή συζήτηση για τα όσα περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο τη ε, συνεργασίας αυτής ε, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και την εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, και εδώ θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής και ας δούμε το τύρι μαντσέγκο ως παράδειγμα, διότι πρόκειται για πολύ σημαντικό προϊόν για το Μεξικό, πολύ σημαντικό προϊόν για την Ισπανία επίσης. Υπάρχει ε, διαφορά μεταξύ του τυριού της Ισπανίας από το τυρί, διότι είναι από πρόβιο γάλα ενώ το τυρί του Μεξικού είναι από γελαδινό γάλα. Στο Μεξικό υπάρχει δυνατότητα να πωλείται ε, τυρί ματσέγκο από την Ισπανία, αλλά και ε, μεξικανικό τυρί ματσέγκο. Αλλά το μεξικανικό τυρί ματσέγκο δεν επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε διαγράμματα ή σχέδια τα οποία να δίνουν μια υπόνοια ότι πρόκειται για ισπανικό τυρί. Ε, αυτό κατά την άποψή μας είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ε, βεβαίως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις γεωγραφικές ενδείξεις που σημαίνει ότι το τυρί Μαντσέγκο το οποίο μπορεί να απολυθεί στην Ευρώπη θα είναι το ισπανικό ε, τυρί με προστασία ονομασίας προέλευσης. Αυτό είναι αυτό το οποίο επιτρέπεται να απολυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για άλλα προϊόντα στις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, στα οποία έχουμε κάνει πολύ σημαντικές ε, συγκεκριμένες προσαρμογές και υπάρχουν και κάποιες ε, ευελιξίες. Είναι πάρα πολύ λίγα τα προϊόντα και θέλουμε να είμαστε απόβλητα βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση για τους καταναλωτές ως προς το ποιο προϊόν αγοράζουν. Επομένως, η επισήμανση όντως είναι πάρα πολύ σημαντική. Και, είμαι στο θέμα της επισήμησης, θα απαντήσω και σε άλλη μια ερώτηση. Το να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την επισήμαση που να είναι πλήρως συμβατά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος να υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα έχουν ετικέτες με τρόπο το, ο οποίος δεν είναι αντίστοιχος με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και όσον αφορά τα μεξικανικά προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να υπάρχει πλήρης ε, ε, σοβασμός ε, των απαιτήσεων της φυτογειονομικής νομοθεσίας. Και βεβαίως η αρχή της προφύλαξης είναι τμήμα του κεφαλαίου των φυτογειονομικών θεμάτων για τις ε, ροές δεδομένων. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πρόσφατα ε, δημοσίευσε την πρότασή της. Αυτή η πρόταση για δεσμεύσεις για τις ροές δεδομένων θα πρέπει ακόμα να συζητηθεί με τα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως ε, δεν υπήρχε χρόνος να παρουσιάσουμε τη νέα πρόταση στο Μεξικό. Υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρηση στη συμφωνία που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε Μόλις είμαστε έτοιμοι με τις εσωτερικές συζητήσεις και έχει τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, να παρουσιάσουμε και την αναθεωρημένη πρότασή μας και να ξεκινήσουμε αντίστοιχες συζητήσεις με το Μεξικό. Αναφέρεται στη συμφωνία εντός ε, διαστήματος τριών ετών, αλλά τίποτα φυσικά δεν μας απαγορεύει να ξεκινήσουμε και νωρίτερα. Όσον αφορά την εφαρμογή, όπως σας είπα και προηγουμένως, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι για να οριστικοποιήσουμε τις συμφωνίες, ε, να γίνει το νομικό χτένισμα και φυσικά πάντα εξαρτάται πόσο χρόνο θα πάρει. Υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις ε, στις οποίες ε, διέρχησε μόνο δύο μήνες. Και από πλευρά Μεξικού είχαμε πολύ κόσμο ο οποίος ασχολήθηκε και με το κείμενο και μπορεί να φτάσει μέχρι και τους έξι μήνες. Εξαρτάται ε, βεβαίω και από τι δύο πλευρέ. Προσπαθούμε και οι δύο να το προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όπω είπα και προηγουμένω, έχουμε και την 1η Ιουλίου εκλογέ στο Μεξικό. Η παρούσα κυβέρνηση ακόμα θα ε, είναι ε, κυβέρνηση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε ολοκληρώσει. Βεβαίως, Δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να περιμένει κανείς ε, να παρουσιάσουμε τη συμφωνία στα κράτη-μέλη πριν ε, το δεύτερο εξάμεινο του 2019 λάβουμε υπόψη και τους χρόνους μετάφρασης και όλες τις υπόλοιπε καθυστερήσεις. Αλλά πάντα φυσικά επιθυμούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Γιατί η νέα κυβέρνηση για το γεγονό ότι τα χέρια του είναι δεμένα. Η νέα συμφωνία δεν θα έχει ακόμα κυρωθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά. Επομένω, η νέα κυβέρνηση ε, θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει. Βέβαια, καλύτερα αυτή η ερώτηση να τεθεί στου Μεξικανού συναδέλφου, αλλά η νέα κυβέρνηση θα είναι αυτή η οποία ε, θα ε, προχωρήσει τη συμφωνία την οποία διαπραγματευθήκαμε. για το αμοιβαίο αποφελέ. Ε, ναι, είναι δύο οι πλευρές οι οποίες διαπραγματεύονται αυτή τη συμφωνία και εμείς από πλευράς μας θεωρούμε ότι είναι υποφελή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι βέβαιη ότι και οι Μεξικανοί συνάδελφοι αντίστοιχα διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία η οποία να είναι προ όφελο και του Μεξικού. Όπω είπα και προηγουμένω. Ο στόχο μια συμφωνία είναι να υπάρχει κάτι το οποίο προσφέρει δυνατότητε και στι δύο πλευρέ να αυξήσουν τι εμπορικέ του συναλλαγές και τι επενδύσει. Υπήρχε και ένα ερώτημα για την κείμενη συμφωνία, η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή. Και αν δείτε τι συνέβη με την κείμενη συμφωνία, το εμπόριο και οι υπηρεσίε τριπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού και είδαμε επίση και μια αύξηση τη τάξη του 7% σε αγαθά σε τήσια βάση που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερη αύξηση από αυτό που έχουμε συνολικά σε άλλες χώρες. Πράγματι λοιπόν ήταν καλές οι εξελίξεις βάσει της παρούσας συμφωνίας, αλλά ε, περιμένουμε τώρα με τις νέες διατάξεις να είναι ακόμα περισσότερο αποφελείς ε, οι εξελίξεις και για τις δύο πλευρές. Αξιολόγηση επιπτώσεων βιωσιμότητα. Ε, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εκ παραλίλου, διότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα η συμφωνία και γιατί βεβαίως ε, επίκυνται εκλογέ ε, στο Μεξικό και υπάρχει ενδιαφέρον να προχωρήσει κάτι εφόσον έχει τεθεί ε, σε κίνηση και επομένως ε, γίνεται ε, και η διαδικασία της εκτίμησης επιπτώσεων. Λάβαμε σχέδια εκθέσεων και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε λάβει υπόψη μια σειρά από θέματα τα οποία τονίστηκαν ιδιαίτερα στο SIA. Ε, δυστυχώς η τελική έκθεση δεν θα είναι διαθέσιμη ε, στην Συμφωνία ε, Εκτίμηση Επιπτώσεων Βιωσιμότητας. Ε, δεν θα έχουμε την έκθεση διαθέσιμη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αλλά φροντίζουμε όσα περιλαμβάνονται σε αυτή την εκτίμηση επιπτώσεων να, έχει ληφθεί, να έχουν ληφθεί υπόψη και στη Συμφωνία. Όσον αφορά την οριστικοποίηση της Συμφωνίας και το τελικό κείμενο, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση για εκρεμή θέματα. Θέλουμε να έχουμε πολιτική συμφωνία για τεχνικές ε, λεπτομέρειες ε, διατυπωμένε με νομικούς όρους. Ε, και αυτό φυσικά προϋποθέτει και κάποιο χρόνο και φυσικά ε, πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με τα προγράμματα. Είναι ε, εκατοντάδες σελίδες, πρέπει να έχουν τη σωστή μορφή και αυτό καθυστερεί. Αυτό αφορά και τις δύο υπηρεσίες και για την πρόσβαση στην αγορά. Θα καθυστερήσει λοιπόν λίγο, αλλά δε, όπως είπα και προηγουμένως δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι υποσυζήτηση, το οποίο να ανατρέψει ε, και να γυρίσει την πλάστικα ή να ε, διαστρεβλώσει τη συμφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για τη Σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δεν υπάρχει καμία απέτηση να εγκριθεί η Σύμβαση 98 σε αυτή τη συμφωνία όπως γίνεται συνήθως και στις προηγούμενες μας συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει καλή συζήτηση με τους Μεξικανούς συναδέλφους και φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις ε, για τη συζήτηση η οποία κρεμεί ακόμα στη Γερουσία στο Μεξικό. το διεθνές ε, δικαστικό σύστημα. Νομίζω ότι τα βασικά στοιχεία του διεθνούς δικαστικού συστήματος, ε, ε, είναι αυτά τα οποία έχουμε στη ΣΕΤΑ. Νομίζω ότι έγιναν αλλαγές στο σύστημα επίλυσης διαφορών στη ΣΕΤΑ από την αρχική συμφωνία και αυτές οι αλλαγές ούτως ή άλλως αντανακλώνται στη Συμφωνία του Μεξικού και Είμαστε βέβαιοι και πολύ ικανοποιημένοι διότι έχουμε μια καλή και στέρεα ε, δέσμευση για το διεθνές ε, σύστημα ε, δικαστηρίων και να υπάρχει ένα πολυμερές σύστημα δικαστηρίων. Για το ξέπλυμα χρήματος και τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα για την καταπολέμηση της ε, διαφοδοράς. Πράγματι και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όσον αφορά την εφαρμογή, όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, μας ενδιαφέρει να γίνεται διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, να υπάρχουν εκθέσεις, να υπάρχει συνεργασία, αλλά ε, όσον αφορά κυρώσεις και επιβολή, κοιτάμε τι γίνεται στο ιστορικό σύστημα της κάθε πλευράς και μετά το ε, συνδέουμε με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί και από το Μεξικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δημιουργούμε ένα ξεχωριστό σύστημα για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ε, υπάρχει και προβλέπεται σε διεθνές πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτά ε, είναι κατά βάση. Όπως σας είπα, όλα αυτά θα ε, παρουσιαστούν ως μία συμφωνία. Είναι μία πλήρη συμφωνία σύνδεσης για την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν δεσμεύσεις στο κεφάλαιο το πολιτικό, ε, ισχυρή δέσμευση μάλιστα για θέματα φύλου και επίσης υπάρχει και μία σειρά ε, προγραμμάτων, 11 τον αριθμό για την ισότητα των φύλων, ε, τα οποία θα προχωρήσουμε ε, και στη συνέχεια. Και φυσικά τα θέματα του φύλου μπορούν να προσθεθούν και στο κεφάλαιο TST που έχουμε και ένα κεφάλαιο για την έλλειψη διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Τώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα υπάρχει σχέση, υπάρχει συμφωνία σύνδεσης ούτως ή άλλως. Ε, υπάρχει σχέση λοιπόν με την βασική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πολιτικό σκέλος. Υπάρχει ενισχυμένο πολιτικός διάλογος και συνεργασία, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και επίσης αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε πέντε συγκεκριμένου τομείς ε, πρόληψη ε, και καταπολέμηση των βασανισμών, ε, εξαφανίσεις, περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους, ανθρώπινα δικαιώματα και έφηβοι και ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις. Αυτά είναι κάτι τα οποία θα προχωρήσουν σε πολιτική σκοπιά και έχουν ενισχυθεί πράγματι στο πολιτικό σκέλος της Συμφωνίας Σύνδεσης. Με αυτό νομίζω ότι ή μάλλον ελπίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλιώς είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω και διμερώς σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κένη. Φυσικά και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, βάλουν υπόψη, ή θέλουν να ακούσουν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζουμε να τη λάβουν και υπόψη και θα επανέλθουμε κυρίως μετά την κακή εμπειρία της Κορέας και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη συμφωνία. Και υπάρχει και η ερώτηση για τη ροή δεδομένων που έχει να κάνει με τόσες πολλές ε, ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις δεν έχουμε πάρει ξεκαθαρή απάντηση για αυτή τη ροή δεδομένων και πώς προστατεύεται. Από την άλλη βέβαια, 21 Μαΐου αρχίζει να ισχύει ο νέος κανονισμός για την προστασία δεδομένων, οπότε θα τα δούμε και υπό το νέο αυτό φως. Ωραία. Ολοκληρώνουμε γι' αυτό, μια που η συγγήτρια έτσι καλώς δεν είναι εδώ για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Όπως είπε και ο πρέσβης, έχουμε αντιπροσωπεία που θα πάει τον Ιούνιο Οπότε θα επανέλθουμε σύντομα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται το σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 4 στην Ευρωπαϊκή στην ημερήσια διάταξη γνώμη έχει να κάνει επίσης με τη Λατινική Αμερική, με τη Mercosur. Και έχουμε εδώ εκπροσώπους ε, πρεσβείας Mercosur. Πρόκειται για την αυτού εξοχότητά του κύριο Γκάουτο Βίλμαν, που είναι πρέσβης της Παραγουάης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον έχουμε εδώ μαζί μας. Και έχουμε και την Σάντρα Γαλίνα, που τη γνωρίζουμε πια καλά, η οποία θα μας παρουσιάσει την κατάσταση πραγμάτων των διαπραγματεύσεων. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Και ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε για να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία δεδομένα της συμφωνίας αυτής. Όπως γνωρίζετε, φτάνουμε στα τελευταία στάδια, ελπίζουμε τουλάχιστον. Τα ζητήματα είναι αρκετά δύσκολα, συνεπώς. Και ουσιαστικά, το τελευταίο γύρο τον είχαμε στην Ασουνσιόν τον Φεβρουάριο. 2 Μαρτίου ολοκληρώθηκε. Είχαμε συναντήσεις, έκτοτε επαφές που ήταν ε, αφοσιωμένες στα πιο δύσκολα ζητήματα. Το καλύτερο σήμερα νομίζω είναι να ακούσω τις ερωτήσεις σας, γιατί είναι περισσότερο ε, να δούμε τι θέλετε να γνωρίζετε και να σας απαντήσω. Χαίρομαι που είναι εδώ και πρέσβης ο Ριγκομπέρτο τον βλέπω, ο πρέσβης της Παραγουάη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και αυτός εδώ, οπότε ίσως και εκείνος πάρει το λόγο. Πρόεδρος, Σέντρα, με εκπλήσει σήμερα. Απίστευτο. Είναι, από σένα ποτέ δεν έχω ακούσει τόσο σύντομη παρέμβαση. Λοιπόν, ωραία. Τότε ο Ιγνάσιο Αλαφράγκα που είναι ο μόνιμο εισηγητής μα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι μόλις έφτασα μετά από ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ και δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω την επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματευτές της Επιτροπής είχαν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αν δεν απατώμε, μπορεί και να απατώμε να με απατάει μνήμη μου, από τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων σε υπουργικό επίπεδο του Δεκεμβρίου στον Πένο, Άιρες, όπου ήταν και ο ΠΟΕ, δεν έχουμε πάρει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Πέρασε δηλαδή ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος. Είμαστε στα μέσα Μαΐου και παρόλο που είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την Επίτροπο, με τις υπηρεσίες σας και με την επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και επιθυμητό να γνωρίζουμε σε τι σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αυτές. Εξάλλου, Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, στην ομιλία του για την κατάσταση πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε σαν στόχο να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Οπότε συμφωνώ με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές και επί τη ευκαιρία της εκθεσής Λόπες και σε άλλες ευκαιρίες. Αυτό ακριβώς εκφράσαμε ως επιθυμία. Αλλιώς θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν έχουμε νέα οι δύο πλευρές ρίχνουν η μία την ευθύνη στην άλλη. Εγώ εδώ καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι για να κάνω κριτική, να τα βάλω με τις χώρες της Μερκοσούρ, αλλά τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές εδώ είμαστε για να προβαίνουμε σε δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Σίγουρα η αρμόδια για τα εμπορικά ζητήματα έχει όλη την καλή θέληση, αλλά προφανώς υπήρξε περιορισμός για κάποια ευαίσθητα προϊόντα. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί, οι βάσεις των διαπραγματεύσεων ήταν ότι έπρεπε να βελτιωθούν οι προσφορές τότε που διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις. Και κάτι άλλο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει τις αρχές της στο ελεύθερο ε, εμπόριο. Λέμε ότι το εμπόριο είναι πρόοδος, είναι ειρήνη, όμως όταν οι εταίροι μας είναι ανταγωνιστικοί, εμείς καμιά φορά τους κλείνουμε τις αγορές μας. Τώρα λοιπόν είμαστε σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσει επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα που είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ε, τοποθεσίε προέλευση και ονομασίε προέλευση και άλλοι ευαίσθητοι τομεί όπω είναι ο πρωτογενή. Δεν πρέπει να χάνουμε πολύ χρόνο, Πρόεδρε, για να δούμε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά να προσπαθήσουμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας και πάλι για να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις. Γιατί ο χρόνος περνάει. Ομολογώ ότι και εγώ έχω κουραστεί λίγο να ακούω και να λέμε ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και πρέπει ήρεμα να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ναι, εντάξει, αλλά απ' την άλλη τρέχει ο χρόνος. Είχαμε στην Παραγουά εκλογέ, τον Οκτώβριο στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στη συνέχεια και μετά έχουμε και τις ευρωεκλογέ. Οπότε, Πρόεδρε, είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή που δεν πρέπει να χάσουμε. Ζούμε σε καιρού με προστατευτικές ε, τάσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Έχουμε και ακρόαση με την ε, ΑΦΕΤ για τη σχέση μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε, τις εμπορικές. Οπότε ζητάω από τους φίλους από τη Μερκοσούρ να είναι ρεαλιστές όσον αφορά τις προθεσμίες για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυτοκινητοβιομηχανία και όλοι να φροντίσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Εγώ ευχαριστώ. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στους και οδησίγητες και μετά έχουν ζητήσει και άλλοι συνάδελφοι. Να βάλουμε χρόνο. Ένα δίλεπτο νομίζω θα είναι καλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και γιατί έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εμπορική συμφωνία υποσυζήτηση. Συνήθως λέμε ότι στο 90% του χρόνου γίνεται το 10% της δουλειάς και στο 10% που εκρεμεί στο τέλος γίνεται το 90% της δουλειάς και χάνεται το 90% των στόχων. Εδώ δίνεται εντύπωση ότι έγινε εξαιρετική δουλειά, στο 10% του χρόνου επιτεύχθησαν κάποιοι στόχοι και μετά ξαφνικά σταματήσαμε. Παύση. Λες και φοβόμαστε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση. Λες και φοβόμαστε να φτάσουμε στην ουσία. Και φάνηκε ότι αυτά ήταν στοιχεία τα οποία αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορούσε ε, την εθανόλη, το ε, βόλιο κρέας και τελικά ε, καταλήξαμε σε αυτά τα σημαντικά θέματα και παρόλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία το είχαμε θέσει επιτάπητος μου φαίνεται ότι δεν έχουν απαντηθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για πολιτικό πρόβλημα και το λέω και στην επικεφαλή των διαπραγματεύσεων για να κατανοήσουμε κατά πόσον η πολιτική κατάσταση στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κυρίως η κατάσταση στη Βραζιλία, οι πρόσφατες εκλογές στην Παραγουάη, που νομίζω δεν ήταν και πρόβλημα, αλλά και η κατάσταση της Αργεντινής, την οποία ε, είδαμε αυτές τις μέρες, η οποία πιέ, ε, ότι πιέζεται διεθνώς για την ε, χρηματοπιστωτική της κατάσταση. Αν αυτά τα στοιχεία λοιπόν σήμερα αποτελούν κόλλημα και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η πολιτική κατάσταση, πρέπει να το δούμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να μου απαντήσει επικεφαλής των διαπραγματεύσεων αν όντω ε, τώρα απλώ ασχολούμαστε με τις τελευταίε τεχνικές λεπτομέρειες ή αν πρόκειται για μια πολιτική παύση. Και θα ήθελα να σταθώ τώρα και σε τρία σημεία στα οποία νομίζω ότι ε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχά, γεωγραφικέ ενδείξει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιε γεωγραφικέ ενδείξει οι οποίε ε, ε, Έχουν κάποιες αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τις ονομασίες. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτά, τι προβλήματα πρέπει να επιλύσουμε σε αυτό το σημαντικό θέμα εμείς ως Ευρωπαίοι, αλλά και οι ίδιες οι χώρες του Μερκοσούρ. Δεύτερον, αρχή της προφύλαξης. Διαβάζουμε στον τύπο κατηγορίες του Υπουργείου Γεωργίας ε, της Βραζιλίας, του Μάτζη, ο οποίος ε, στην ουσία κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρησιμοποιεί φυτογειονομικές ε, προφάσεις ε, για λόγους προστατευτισμού. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να πούμε τα πράγματα στα ράτα. Πρέπει να κάνουμε τη συμφωνία, αλλά όχι και να υπαναχωρήσουμε σε αρχές που αφορούν τα φυτογειονομικά ζητήματα, όπως σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Και τέλος, κάτι τελευταίο, το θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Ε, κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα. Έγιναν πολλές συναντήσεις εδώ στις Βρυξέλλες με την κοινωνία των πολιτών, η οποία μας επισημαίνει ότι το επίπεδο ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών ε, στις χώρες του Μερκοσούρ δεν είναι τόσο υψηλό. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να φροντίσει και αυτό το, το σκέλος να τεθεί ε, υπόψη ε, των συνομιλητών μας. Εγώ εξακολουθώ να αισιοδοξιώ. Είναι αισιοδοξία όμως γιατί θέλω να το επιτύχουμε και δεν ξέρω αν θα το επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταμπάν. Θα ήθελα να πω και εγώ το εξής. Μπορεί να κλείσει για πολλούς λόγους αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε, όπως λέγεται. Και μπορεί η περίοδος του ελευθέρου εμπορίου σιγά σιγά αναπνέει τα λίστια. Αν κοιτάξουμε τι μας επιφυλάξουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία με τη μέρκοσού. Μερικά κρίσιμα σημεία. Ασκούσαμε για την αυτοκινητοβιομηχανία 40%, ε, 45% είναι θέματα ποσοστώσεων εκεί ενδιαφέρονται οι χώρες Μερκοσούρ όσο γίνεται να έχουν δική τους παραγωγή. Αλλά αυτό το θέμα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κανονικά δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα. Εγώ είμαι οικονομολόγος και καταλαβαίνω ότι όταν κάπου μπλοκάρεται κάτι ε, σημαίνει ότι θέλεις ανταλλάγματα. Και για την αυτοκινητοβιομηχανία πραγματικά το έχουν στυλώσει εκεί. Τι θέλουνε οι Μεξικανοί, λέει ο κύριο Σταρμπάτη, σε αντάλλαγμα. Το μέγα πρόβλημα είναι το εμπόριο με τα γεωργικά προϊόντα. Το έχω ζήσει κάθε φορά που πάω στη Λατινική Αμερική. Τι κάνετε εκεί στις διαπραγματεύσεις και θέλω να καλέσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχωρήσει λίγο. Γιατί όταν έχουμε περισσότερες εισαγωγές από τις χώρες Σουρ, αυτό είναι καλό και για τους καταναλωτές μας. Τι μανία έχουμε να σκεφτόμαστε μόνο τους παραγωγούς, να σκεφτούμε λίγο και τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Εντάξει, έχουμε αγρότες, έχουμε και καταναλωτές όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή, για να μην πω η σημαντικότερη. Και ε, θα αφήσει και εποχή για το ελεύθερο εμπόριο. Το καταλαβαίνουν αυτό. Οι διαπραγματευτές ξέρουν τι τους περιμένει και τι ευθύνη έχουν. Έχουν καταλήξει τι θα κάνουν απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αν μπλοκάρουν και άλλα ρεύματα εκτός από το αλουμίνιο και το χάλιβα. Βασικά ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται και ευαγγελίζεται την προστασία της Αμερικανικής βιομηχανίας. Θα πρέπει και εμείς να στείλουμε ένα μήνυμα υπέρ του ελευθέρου εμπορίου και κατά του προστατευτισμού. Αυτός είναι ο προορισμός μας πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ε, αναλάβουμε τις ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Η Τίτα Χαράνσοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Είναι λίγο απίστευτο αυτό, γιατί μόλις ε, τελειώσαμε τη συζήτηση για τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Ελευθερίου Εμπορίου με το Μεξικό και τώρα συζητούμε αυτό. Αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε με το Μερκοσούρ το 1999 ένα χρόνο πριν τη θέση σε ισχύ της ελεύθερη συμφωνίας με το Μεξικό. Πραγματικά τελειώνει ο χρόνος. Όλο λέμε για ευκαιρία και παράθυρα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αιώνιο αυτό. Ακούμε διάφορες προθεσμίες που αλλάζουν. Στην αρχή μας είπαν το Γενάρη, μετά τέλη Μαρτίου, μετά Ιούλιο. Ας είμαστε ειλικρινείς όμως υπάρχει κανένα πραγματικό χρονοδιάγραμμα για μας, για το πότε θα σταματήσουμε. Και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Για την αυτοκινητοβιομηχανία διαβάσουμε πολλά δημοσιεύματα πρόσφατα στον, κήπο, στον τύπο. Συγγνώμη. Και επειδή είναι τόσο σημαντική η αυτοκινητοβιομηχανία για την Ευρώπη, θέλω να ακούσω περισσότερα από την κυρία Γκαλίνα. Τι συμβαίνει πραγματικά στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Από τους πρασίνους. Ο Γιάννη Ξαντώ, αγαπητός μου αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γεγονό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν μας λέει και πάρα πολλά για το τι συμβαίνει πραγματικά στις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω στις απαντήσεις να μάθουμε περισσότερα. Αλλιώς θα συζητάμε μεταξύ μας και εσεί θα είστε παρατηρήτρια. Αλλά τι νόημα έχει να σα δίνουμε το λόγο και με το συμπάθειο κιόλα, αν δεν μαθαίνουμε και πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφο Ντάντι αναφέρθηκε στην αρχή τη προφύλαξη. Υπάρχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, ε, κατά τις αρχές προφύλαξης. Πώς το λαμβάνετε αυτό υπόψη στην σημερινή κατάσταση των διαπραγματεύσεων και που βρίσκονται γιατί γνωρίζουμε ότι το 100% σχεδόν τη σόγιας που εξάγει η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι μεταλλαγμένη. Και πώς θα κάνουμε δοκιμές για να δούμε το ποσοστό. Το, το θέμα της γλυφοσάτης που είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και το θέμα της υγείας γενικότερα. Γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν τρομακτικά σκάνδαλα εκεί, ε, υγειονομικά, στο κρέας, ειδικά στη Βραζιλία και πάλι. Και τέλος, εντάξει, εγώ ακούω ξανά και ξανά ότι η Ευρώπη θέλει να αντισταθεί κατά της απορρίθμισης του κλίματος και να προστατεύει την δημόσια υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και να προστατεύει και τους αγρότες. Μα αν υπάρχει μία συμφωνία που καταστρέφει τον Αμαζόνιο είναι τούτη εδώ, με τις εξαγωγές αυτές. Ε, βοηού κρέατος κυρίως. Και ξέρουμε ότι μηχανικά για κάθε σφάγιο βόιο που εξάγεται πόσα δέντρα καταστρέφονται στον Αμαζόνιο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο. Και μετά ε, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ε, αναφέρθηκε και ένα ε, δευτερεύον και σχετικό ερώτημα για τις υπηρεσίες. Η ε, Ουρουγουάη και η Παραγουάη κατέληψαν τις διαπραγματεύσεις της για τις υπηρεσίες. Τι γίνεται με αυτές. Και ένα τελευταίο που συνδέεται και με την αρχή της προφύλαξης. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ξέρετε πόσο ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να μην είναι ε, έτσι, διακοσμητικό ε, το κεφάλαιο αυτό από πλευράς επιβολής κυρώσεων. Και ο πρόεδρος Λάγκε ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό και το παρακολουθεί και εμείς επίσης. Τι θα γίνει, θα κινηθούμε καθόλου ευκεί, σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Μέρκοσουρ από την Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Χελμουτσόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σάντρα Γκαλίνα ε, ε, που παρακολουθεί μόνιμα ε, την ομάδα παρακολούθησης ΙΝΤΑ τη συμφωνία με το Μερκοσούρ, γιατί το Κοινοβούλιο δεν κάνει τι διαπραγματεύσει, αλλά τι παρακολουθεί και τι ελέγχει με επικριτικό μάτι και τελικά θα πρέπει να δώσει τη συνένεση του ή να μην τη δώσει τη σύμφωνη γνώμη το Κοινοβούλιο. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Πριν από δέκα μέρες ως πολιτική ομάδα είχαμε μια πολύ μεγάλη διάσκεψη ε, για τι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωση Μερκοσούρ για την εμπορική συμφωνία εδώ, στο Κοινοβούλιο και ήταν παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ ρητά για την παρουσία τη. Αλλά οι δηλώσει ήταν αρκετά αντιφατικές. Είχαμε πολλούς εκπροσώπους από την πολιτική, από την κοινοβουλευτική δομή, από την κοινωνία των πολιτών και από τις χώρες Μερκοσούρ και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα θέματα των φυτοφαρμάκων στη Βραζιλία, ας πούμε, και η προστασία του περιβάλλοντος, η Γεωργία ήταν ζήτημα. Η επιστηστική ασφάλεια, πολύ μεγάλο θέμα. Είχαμε εκπροσώπους του Food Watch, οι οποίοι κατά την άποψή μου και δικαιολογημένα ε, φώτισαν κρίσιμες πτυχές που έχουν σχέση ε, και θα τα βρούμε μπροστά μας με τη Συμφωνία Μερκοσούρ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δύο μηνύματα γιατί δεν έχουμε και χρόνο για να κάνουμε μεγάλες συζητήσεις σήμερα. Πώς έχει η πολιτική κατάσταση στο σύνολό της και ευχαριστώ τους εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος που είναι παρόντες από τις χώρες Μερκοσούρ θα πρέπει να είναι δύσκολο να πορευθούμε, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα πολιτική σε πολλές χώρες, ήδη αναφέρθηκαν Βραζιλία και Αργεντινή. Πώς μπορούμε σοβαρά να βάλουμε ένα χρονικό όριο μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τον Νοέμβριο. Ε, μια εμπορική συμφωνία έχει λιγότερο σχέση με το ελεύθερο εμπόριο και περισσότερο με το δίκαιο εμπόριο. Και εκεί θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται όλα τα θεμητά συμφέροντα των πολιτών. Δηλαδή πώς με τις εμπορικές σχέσεις θα βοηθήσουμε ε, να προχωρήσει η κοινωνία ε, στις χώρες αυτές. Αλλιώς ε, θα μας αφαιρέσουν την εμπιστοσύνη οι πολίτες και αφορά και εμάς και τις χώρες εταίρους στην Αμερική. Λοιπόν, για την αρχή της προφύλαξης και όλες αυτές τις αρχές που αναφέρθηκαν πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη και να τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι οι οποιασδήποτε προστατευτικές τάσεις ή πειρασμοί, αλλά ε, μια εμπορική συμφωνία προς όφελος των λαών και του περιβάλλοντος φυσικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατο. Όχι κύριε Ντάτμουθ, η κυρία Μπεγκίν είναι σκιώδη εισηγήτρια πρώτα. Ε, Αλλά είναι από την ομάδα σας αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, χρειάζομαι και το μικρόφωνο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλά και για τη θέση μας. Νομίζω ότι εμείς θεωρούμε ότι σε αυτές τις ε, τελικές διαπραγματεύσεις, καλό είναι να επαγρυπνούμε για κάποια σημεία της συμφωνίας, όπως για παράδειγμα τον κίνδυνο να έχουμε πολύ ε, αυξημένο αριθμό εισαγωγών ε, βόηου κρέατος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους ε, παραγωγούς. Ούτως ή άλλως οι κτηνοτρόφοι μας οδηγούν σε αυτάρκεια στην παραγωγή του βόηου κρέατος, επομένως θα έπρεπε να περιορίσουμε τις αγωγές στο θέμα αυτό. Επίσης, μας ανησυχεί ιδιαίτερα και το θέμα των διατροφικών μας προτύπων, τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν κινδύνο με αυτή τη συμφωνία για να μην αναφέρω και πιέσεις σε ζώα και περιβάλλον. Ε, κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί, η πιθανή εισαγωγή πολύ μεγάλων ποσοτών βιοκαυσίμων στην Ευρώπη που μπορεί να είναι εις βάρος του περιβάλλοντος. Ε, ε, ο συνάδελφος Σούλτς αναφέρθηκε και στην όλη διαδικασία. Δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αντίκτυπο στη συμφωνία. Για παράδειγμα, στη Βραζιλία, μήπως η νέα κυβέρνηση ε, δεν θα έχει αρκετή ευελιξία για να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου οι συζητήσεις ακόμα δεν είναι ικανοποιητικέ ε, για τους ε, παραγωγούς μας. Και επίσης το μόνο πλεονέκτημα θα μπορούσε να είναι από γεωργική σκοπιά αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της αμοιβαιότητας. Για παράδειγμα, στο εμπόριο των ίνων. Το θέμα είναι απλό. Το ευρωπαϊκό ε, κρασί πληρώνει 20% ε, φόρους, ενώ εμείς ε, χρεώνουμε 10% δασμούς για την εισαγωγή των δικών τους τους κρασιών. Και υπάρχει και θέμα για τις δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε περισσότερους διαγωνισμούς. Και μία ερώτηση. Όσον αφορά το εμπόριο ζάχαρης από ζαχαρότεφυλα, θα μειωθεί... Ο ζαχαροκάλαμο, συγγνώμη, θα μειωθεί ο δασμός ε, για την εισαγωγή και αν μια αντίστοιχη συμφωνία με αυτή του Μεξικού θα επιτρέψει να επιταχύνουμε τη διαδικασία στο Μερκοσούρ και σε ποιο τομέα. Ευχαριστώ. Και τώρα για το ENF, η κυρία Ζαμέ, κάθεστε δίπλα. Ε, τι έχετε, νέα <laughs> συμμαχία, νέο συνασπισμό. Όχι, όχι. Ελπίζω, ελπίζω. Άκουσα του συναδέλφους να αναφέρονται σε πλεονήματα για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να πω εδώ ότι η κατανάλωση ε, κρέατος μειώθηκε κατά 27% Απειλούνται λοιπόν ε, θέσεις εργασίας ε, ε, κυρίως στον τομέα του βόλου και φυσικά με εισαγωγές από τον Καναδά, από το Μερκοσούρ. Να υπενθυμίσω ότι πάνω από το μισό της ευρωπαϊκής παραγωγής εισάγουν. Επομένως δεν είναι θέμα προστατευτισμού, πρέπει να σώσουμε τους παραγωγούς μας. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για προστατευτισμό και κύριε Ζαντώ αναφερθήκατε στο νερό και συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει, συμμαχία μέχρι εκεί ο κύριος Νταντάν λοιπόν επέστρεψε από μία αποστολή μελέτης και διαπίστωσε ότι υπάρχουν σκάνδαλα σε θέματα υγείας και κρέατος. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν ουσίες οι οποίες απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρόκειται λοιπόν για μέτρα προστατευτισμού για του καταναλωτέ μα και δεν λαμβάνονται υπόψη. Ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την ειχνηλασιμότητα και τι ε, επισημάνσεις και θα ήθελα να ρωτήσω και πάλι τι κάνουμε για του καταναλωτέ, πώ του προστατεύουμε του καταναλωτέ, και πραγματικά θεωρώ ότι αυτά είναι ουσιαστικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων για τα οποία ε, υπενθυμίζω ότι είμαστε αναφανδόν κατά αλλά επίσης ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και πάρα πολύ καλά του καταναλωτέ μα ενδιαφέροντες ε, οι καιροί συμμαχίες, ε, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά και πρασίνους, ε, τέλος πάντων. Ο Ντέιβιτ Μάρτιν στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι ετέθησαν μέχρι τώρα. Καταρχάς πρόσβαση σε φάρμακα. Πάντα στις συμφωνίες προσπαθούμε να έχουμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ να υπάρχει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για τις επιχειρήσεις μας, αλλά να μην περιορίζεται η πρόσβαση στα φάρμακα. Η Βραζιλία είναι ένα από τα εργαστήρια γενώσιμων φαρμάκων του κόσμου και είναι πολύ σημαντικό η Βραζιλία να μπορεί να απολύει ε, τα προϊόντα της, ε, τα γενώσιμα παγκοσμίω γιατί βοηθά ε, σε όλο τον κόσμο. Έχω... διασφάλιση από τη Σάντρα ήδη ότι προσπαθούμε να το λάβουμε επίσης του και επίσης τι γίνεται με τις συμφωνίες TRIPS ε, ε, συν σε κάποιες χώρες και πώς δυσχεραίνει αυτό τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερη ερώτηση, ακόμα πιο ε, σύντομη. Ξέρουμε ότι το Μεξικό προχωρήσαμε τα πράγματα, έχουμε τη συζήτηση και έχουμε και έναν από τους καινοτόμους παράγοντες της Συμφωνίας του Μεξικού για την ευημερία των ζώων. Θα έχουμε αντίστοιχο κεφάλαιο για την ευημερία των ζώων και στη Συμφωνία για το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ. Η Καρολίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από κανένα δύο εβδομάδες ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους μικρούς γεωργούς στη Βραζιλία. Με ανησυχούσε το θέμα, δεν μου απάντησαν. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω και την ερώτηση προφορικά. Μήπως η συμφωνία του Μερκοσούρ θα μπορούσε να, πλέξει, να πλήξει πολύ σοβαρά τους ε, μικρούς γεωργούς. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερα φυτοφάρμακα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι και ε, τα δάση του Αμαζονίου κόβονται και ε, αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκοπεύετε να κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτές τις εξελίξεις και ε, αν υπάρχουν προβλέψεις για κυρώσεις στο κεφάλαιο της βιωσιμότητας. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες κυρώσεις όταν υπάρχουν παραβιάσεις και γιατί ε, είναι η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος μια ερώτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προβλέπεται να υπάρχει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί η κατάσταση σε πολλές χώρες της Μερκοσού είναι ιδιαίτερως ανησυχητική. Για παράδειγμα, ε, εκδίωξη ανθρώπων από τη γη τους. Μήπως αυτοί ε, οι παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα οδηγήσουν σε ενεργοποίηση της ρήτρα και αν δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει. Ε, η αρχή ενεργοποίησης ρήτρα δεν είναι εύκολη απάντηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Ιάν Μινέρ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα την κυρία Σάντρα Γαλίνα. Ήλπιζα ότι θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η συμφωνία. Δεν το έκανε όμως, δυστυχώς. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι γίνεται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριο Χόγκαν έχει μιλήσει ε, για την ε, συμφωνία και ακούσουμε και από, για τη Βραζιλία πράγματα, αλλά δεν υπάρχει καμία σαφήνεια. Γι' αυτό θα ήθελα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα θέλαμε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να απαντήσει στην κριτική που ακούγεται. Τι γίνεται με τη γεωργία, με το περιβάλλον, για τα φάρμακα ρώτησε ο Ντέβιτ Μάρτιν, οι οικονομικές ροές. Όλα αυτά παραμένουν σε κρεμότητα και δεν αποτελεί έκπληξη και δεν είναι εξαίρεση η συμφωνία αυτή με τη Μερικοσούρ... Έπειτα, ε, όταν γίνονται παρεμβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει διαφθορά, όλα αυτά περνάνε ατιμωρητή. Ε, αυτή η κριτική ακούγεται. Πώ αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώ τη λαμβάνει υπόψη στι διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις εν ώψη τη συμφωνίας. Ευχαριστούμε. τελευταίο, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό βέβαια. Παρακαλώ, ναι, εγώ να συγχαρώ την Μερκοσούρ που το 2016 απέκλεισε τη Βενεζουέλα. Αν και άλλες χώρες είχαν ε, τοποθετηθεί με τον ίδιο τρόπο, αυτό θα βοηθούσε πολύ και το, οι εργατικοί, αν το είχαν κάνει. Τώρα η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Έτσι, έτσι δεν προτάθηκε. Ναι, ωραία γνέφει ε, καταφατικά η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Μία ερώτηση έχω λοιπόν προς την Επιτροπή. Εφόσον είναι ελεύθερων συναλλαγών, εσείς προτείνετε ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, έχετε τέτοια ρήτρα και αν όχι, γιατί όχι. Και για τις θεωρήσεις, τι προτείνετε. Χαλάρωση των απαιτήσεων, αλλά η κύρια ερώτησή μου είναι υπάρχει ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας. Και αν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει, γιατί επιμένει για την ελεύθερη κυκλοφορία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλου είδους συμφωνίες και θέλει να την επιβάλλει την ελεύθερη κυκλοφορία. Πρόεδρος, ωραία. Ο κύριος Κάτω φύρμα τώρα πρέσβης. Αλλά να προσθέσω προηγουμένως μια ακόμα ερώτηση κι εγώ. Άκουσα με Σάντρα. Βεβαίως, οι διαπραγματεύσει λαμβάνουν χώρα την ίδια εποχή που συζητάμε και τον Brexit, ναι. Τι προβληματισμός υπάρχει σε μια τέτοια συμφωνία εν ώψη του Brexit. Επηρεάζει το Brexit. Δηλαδή θα μπορούσε να προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο και η διαπραγμάτευση για το Brexit. Είναι μια γενική ερώτηση, έτσι, για τις διαπραγματεύσεις μας. Ωραία, ο κύριος Βήμαρ. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να σας πω ότι για μας, τους εκπροσώπους της Μερικοσούρ, είναι μεγάλη ικανοποίηση αλλά και προνόμιο που μας δίνεται την ευκαιρία να απευθυνθούμε στους αξιότιμους ευρωβουλευτές της Επιτροπής αυτής Διεθνούς Εμπορίου. Πιστεύω πραγματικά, όπως το ακούσαμε ήδη, ότι έχουμε φτάσει στο πιο περίπλοκο στάδιο των διαπραγματεύσεων, με πιο ευαίσθητα ζητήματα. Τώρα τίθεται τα πιο δύσκολα θέματα. Έχουμε διανύσει βέβαια μεγάλο δρόμο για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Και τώρα μένει να λυθούν τα τελευταία προβλήματα, τα δύσκολα. Οπότε ίσως δεν είναι η στιγμή για να συζητάμε για επιμέρους θέματα. Αυτό όμω στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι η Μερκοσούρ έχει αναλάβει την υποχρέωση σε ανώτατο επίπεδο να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Έχουμε συχνά συναντήσεις, βίντεο διασκέψεις ανάμεσα στους δικούς μας συμβούλους, επιτετραμένους, υπουργούς, αρμόδιους για το εμπόριο, προκειμένου να έχουν οι διαπραγματεύτες μας την κατάλληλη στήριξη και την απαιτούμενη στήριξη. Αυτό έχει αποφασιστεί. Όπως επίσης διευκολύνεται η έλευση εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες, όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι η Μερκοσούρ είναι ενωμένη και από κοινού διαπραγματεύεται βάσει στόχων και βάσει προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στις διαπραγματεύσεις αυτές από το πρώτο στάδιο τους. Επίσης, η Μερκοσούρ, πρόεδρε, είναι πολύ προσεκτική για να αποφύγει το blame game, δηλαδή να τα ρίχνουμε στους άλλους, για να διευκολύνουμε τις επαφές και τις σχέσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Και απευθείας απευθυνόμαστε στους συνομιλητές μας, δεν ε, διαραίουμε πράγματα στον τύπο, μιλούμε με την επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι αποφεύγουμε ο τύπος, τα περιοδικά, εφημερίδες να αναφέρονται στις διαπραγματεύσεις αυτές με απρέπεια. Υπάρχει σαφής βούληση από τις κοινωνίες μας υπέρ της συμφωνίας αυτής. Υπάρχουν ε, βέβαια τομείς που θέλουν να προστατεύσουν ε, τα συμφέροντά τους και υπάρχουν ε, και κάποιες ομάδες που είναι έτσι καλλιώς κατά οποιασδήποτε συμφωνίας. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Πιστέψτε με όμως, υπάρχει ευρία βούληση για να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις εφόσον λυθούν τα πιο δύσκολα ζητήματα. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, Πρόεδρε, ότι οι θυσίε πρέπει να κάνουν και δύο πλευρές. Γιατί δεν θα είναι δυνατόν να έχουμε συμφωνία όπου η μία πλευρά θέλει να προστατεύσει τους ευαίσθητους ε, κλάδους της και να ζητάει άνοιγμα από την άλλη πλευρά υπέρ της. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια από τις δύο πλευρές και από τη Μερκοσούρ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει να γίνουν θυσίες και να αφήσουμε στην πάντα τον προστατευτισμό. Και πρέπει να εγκαταλείψουμε κάθε ιδέα πατερναλισμού. Όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους δικούς μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε δίκαιους κανόνες, όπως το είπαν και εξότιμοι ευρωβουλευτές. Προσπαθούμε να έχουμε όχι μόνο μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αλλά πάνω απ' όλα προσπαθούμε να έχουμε μια δίκαια συμφωνία. Και η Μερκοσούρ έχει δεσμευτεί υπέρ αυτού του στόχου, δηλαδή του να πετύχουμε μια δίκαια συμφωνία. Αυτά είχα να πω σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας και τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για την ευκαιρία που μου δώσετε να απευθυνθώ σε εσά εκ μέρους της Μερκοσούρ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρέσβη. Και τώρα η Σάντρα για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που καλέσατε και τους πρέσβεις. Πολύ χαίρομαι που ακούσαμε τον πρέσβη της Παραγουάης και τα τόσο λογικά που μας είπε, γι' αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουν παρεξηγήσεις ή κάποια πράγματα να μην ξεκαθαριστούν. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης. Δεν πρόκειται μόνο για εμπορική συμφωνία. Και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι υπάρχει μια πολιτική πτυχή σε αυτήν την τεράστια συμφωνία που βέβαια μερικές φορές ε, επικαλύπτεται από αυτά τα οποία έχουμε με το χάλιβα, το αλουμίνιο κλπ. που πάνε βέβαια πέρα από τη συμφωνία αυτή, Ωραία, την επηρεάζουν. Τώρα να απαντήσω πρώτα σε αυτό που ρωτήσατε για το Brexit. Ξέρετε, το Brexit και όλα τα σχετικά, πώς να το πω, επηρεάζουν σε ένα βαθμό όλες τις διαπραγματεύσεις, έχουν κάποιες ε, επιπτώσεις. Ε, κοιτάξτε, δεν μας είναι αδιάφορα και αυτά που γίνονται στην ε, Κίνα με τη, το δικό τους, τις δικές τους ε, εξαγωγές σε εμάς τις υπερβολικές. Όλα αυτά επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις. Δεν είμαστε απομονωμένοι. Συνεπώς, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και το Brexit είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που παρεμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις και όχι το μόνο. Το πρώτο στοιχείο που πάντα εμφανίζεται όταν συζητάμε τέτοιες συμφωνίες είναι η γεωργία. Η γεωργία είναι μια δύσκολη περίπτωση σε αυτή τη συμφωνία, γιατί είμαστε συμπληρωματικοί κατά κάποιο τρόπο. Και εγώ θα ήθελα να σας ε, μεταφέρω ότι είναι σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση ε, αυτού του ζητήματος. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξουν μεγάλα κέρδη για τη γεωργία στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι αλήθεια ότι πρόκειται μόνο για τα γαλακτοκομικά. Όχι. Υπάρχει προστασία των ζώων. Ναι, θα υπάρχουν διατάξεις επ' αυτού. Προσπαθούμε ακόμα να δούμε αν θα είναι κεφάλαιο ή όχι, αλλά θα έχουμε διατάξεις και για την ε, μικροβιακή αντοχή. Οπότε και η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται στο, για τα θέματα αυτά και θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Μην νομίζετε ότι επιμένοντας στα δικά μας θα κερδίσουμε. Όχι. Αν συμφωνήσουμε χωρίς να αλλάξουμε το σύστημά μας έτσι, γιατί η συμφωνία δεν έχει σαν στόχο να αλλάξει το δικό μας σύστημα, θα το διατηρήσουμε. Όμως θα είμαστε πιο δυνατοί θεσμικά ε, σε όλα τα φόρα που θα συζητιούνται αυτά τα ζητήματα. Και έρχομαι και στο δεύτερο που έχουμε κέρδη για την Ευρώπη. Και αυτό είναι ο τομέας υγειονομικός και φυτογειονομικός. Δεν θα πέσουν οι προδιαγραφές μας, όχι. Και στη συμφωνία αυτή, επειδή είμαι πεπισμένη ότι είναι ένα πολύ ε, σοβαρό ζήτημα, δημιουργήσαμε ένα κεφάλαιο το οποίο βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα σημαίνει ότι θα έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές. Δηλαδή, και οι χώρες της Μερκοσούρ θα είναι οι σύμμαχοί μας στον αγώνα αυτά γιατί θα κρατήσουν ψηλές προδιαγραφές. Γίνεται. Εγώ δεν είμαι μόνο υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαι και πολίτης και ε, εκπλήσωμαι μερικές φορές και σοκάρομαι από αυτά που ακούμε. Ε, τα ξαπάτε συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε να γίνονται απάτες, εννοείται, να μην ε, φτάνουν στην αγορά μας, προφανώς. Το κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου, ελπίζω να το διαβάσετε, εκεί θα βρείτε κεφάλαιο για το οποίο είμαι περήφανη για τα φυτογειονομικά. Τώρα για την αρχή της προφύλαξης. Πρέπει να απαντήσω στον αξιότυπο Νταντέ. Στηρίζεται με τους πιο ισχυρούς όρους, θα το δείτε. Υπάρχει και στο TSD, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα που πηγαίνει πέρα από τα φετογειονομικά βέβαια. Και από αυτού να προσθέσω κυρώσεις, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε προτείνει την υλοποίηση, έτσι όπως την προτείνουμε τώρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για ένα σύστημα που θα βελτιώσει την κατάσταση. Και επιτρέψτε μου, ακόμα και αν συζητήθηκε πολύ το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαπραγμάτευση αυτή, είμαι περήφανη που έμεσα οι διαπραγματεύσεις μας προωθούν τη συζήτηση. Και θα έλεγα μάλιστα ότι κάθε φορά που είμαστε στην περιοχή, εγώ για παράδειγμα, ζητάω πάντα ε, να οργανώνονται συναντήσεις με την κοινωνία των ε, ε, πολιτών. Και πρέπει να ευχαριστήσω και τους συνομιλητές μου γιατί φρόντισαν και ήταν και παρόντες αυτές τις συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών. Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς την κοινωνία των πολιτών. Μπορεί να είμαστε καταναλωτές, αλλά δεν είμαστε μόνο καταναλωτές. Πρέπει να κοιτάμε ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπων που έχουμε απέναντί μας. Ελεύθερο εμπόριο, εντάξει, δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε συμφωνία που να προωθεί τις αξίες μας. Μπορεί να διαφέρουμε όσον αφορά τις κυρώσεις με τον πρόεδρο Λάγκε, αλλά εγώ έχω δεσμευτεί για όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά δικαιώματα και για το οποίο νοιάζομαι πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να έχουμε δίκαιο εμπόριο χωρίς να υπάρχει δίκαια μεταχείριση. Τώρα, ανθρώπινα δικαιώματα ρωτήσατε. Ναι, καλύπτονται και υπάρχουν και κυρώσεις. Γιατί ανήκουν στην κατηγορία των βασικών στοιχείων για τα οποία προβλέπονται κυρώσεις. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι για τις βασικές συμβάσεις που περιλαμβάνουμε στο κεφάλαιο TST υπάρχουν και τα δικαιώματα. Τα κέρδη, το φέλη για τη Γεωργία είναι και οι γεωγραφικές ενδείξεις και περισσότερες εξαγωγές προς τις χώρες αυτές. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις είναι κάτι που το συστήνει και η Μερκοσούρ. Καταλαβαίνετε ότι η προοπτική μας είναι τελείως διαφορετική η οπτική γωνία μας. Αλλά τώρα φτάνουμε ε, για κάποιες ονομασίες στη στιγμή της αλήθειας. Και τώρα πρέπει η εταίροι μας, το οποίο πρέσβης της Παραγουάης, να μην αφήσουμε ε, κανέναν να προχωρήσει σε κατάχρηση τέτοιων ονομασιών και να τις χρησιμοποιεί παράνομα. Τώρα θέλω να απαντήσω για το ζήτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί πολλά γράφονται στον τύπο επ' αυτού, εξαιτία της επιρροής ε, αυτού του διδήμου Μεξικό-Μερκοσούρ. Θέλω να διευκρινίσω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές διαπραγματεύσεις. Για το Μεξικό υπήρχε μια ενημέρωση της συμφωνίας, εδώ πέρα είναι κάτι πιο σημαντικό. Ε, το θέμα της προέλευσης. Πολλοί επικεντρώνονται σε αυτό. Πάντως στη Μερκοσούρ πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και διαφορετικές θέσεις, γιατί υπάρχουν χώρες που θα θέλαν τη συνορμολόγηση οχημάτων με ευέλικτους κανόνες και άλλοι που είναι λιγότερο ευέλικτοι γιατί έχουν τις δικές τους ε, αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν να προστατεύσουν. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα για το χρόνο της ελευθέρωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας που δεν ικανοποιεί ακόμα αν και είναι φημισμό το δεν ικανοποιεί ακόμα, τέλο πάντων. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στι ανάγκε μα και τι ανάγκε των εταίρων. Ίσως εξετάσουμε το θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και βάσει του TBT. Ξέρετε ότι θέλαμε ένα παράρτημα, γιατί πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι το πρώτο. Ε, προβάλλουμε την κατάσταση στο μέλλον. Ξέρουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε κάποια στιγμή αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, που θα το οδηγάει η Google, ξέρω εγώ. Οπότε, για το TBT θέλουμε κάτι κατάλληλο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι σημαντική μόνο μία πτυχή για τα αυτοκίνητα, είναι πιο συνολικό το θέμα. Και θα ολοκληρώσω με τα φάρμακα, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτές οι χώρες της Μεσκοσούρ όχι μόνο δεσμεύονται με την συνθήκη για την κλιματική αλλαγή και όλα τα υπόλοιπα. Και εμείς έχουμε υπογράψει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, το 3,8, που λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε την ε, παγκόσμια κάλυψη υγείας. Ξέρω ότι στην Βραζιλία είπαμε ότι θα πρέπει οι θεραπείες να φτάνουν και στους πιο φτωχούς και στις πιο φτωχές χώρες. Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή διατύπωση στο κείμενο αλλά η Ευρώπη θέλει να προστατεύσει το θέμα αυτό των φυτογειονομικών και την υγεία για όλους. Τώρα ζητώ συγγνώμη αν δεν απάντησα σε όλα. Α, για τις υπηρεσίες να πω ακόμα ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε την μετανάστευση και τις υπηρεσίες. Εδώ θα υπάρχει ποσόστοση για εμπειρογνώμονες οι ανθρώπους δηλαδή που έχουν τα προσόντα να ταξιδέψουν. Και αυτό υπάρχει στο κεφάλαιο των υπηρεσιών. Δεν είναι κεφάλαιο για τη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ λοιπόν και συγγνώμη αν δεν κάλυψα όλα τα ζητήματά σας. Πιστεύω όμως ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει να συνεχιστεί με κάποια μορφή. Φυσικά. Έχουμε μια σημαντική ερώτηση διευκρινιστική από τον κύριο Ζαντό για τον Brexit. Υπάρχει ένα ειδικό θέμα που είναι οι ποσοστώσεις ε, και οι δασμοί. Από 70 τόνους βοηού πάμε σε 100.000 τόνους βοηού κρέατος. Και αυτό πώς θα επιμεριστεί ανάμεσα στα εναπομείναντα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί είναι μεγάλη αγορά η Βρετανική. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε. Πώς θα μοιραστεί αν υπάρξει συμφωνία η ποσόστοση του Ηνωμένου Βασιλείου να, να μην καταλήξει στην ευρωπαϊκή αγορά. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά αφορά την ε, υψηλή πολιτική, έτσι, κάποια υψηλά αμοιβόμενα στελέχη. Ξέρουμε ότι επίκειται το Brexit και αυτό δεν αφορά μόνο το βόλιο κρέα, αλλά και άλλα προϊόντα και το έχουμε υπόψη μα. Το βόλιο κρέα είναι ένα μόνο από τα προϊόντα και κατά τα άλλα έχουμε και ποσοστώσεις δασμολογικές. συγκεκριμένες για τα προϊόντα, για τη ζάχαρη, ας πούμε, για το βόλιο κρέας και για άλλα. Δεν είναι κάτι έτσι γενικό και όριστο. Υπάρχουν και πολύ ευαίσθητα προϊόντα φυσικά έχουμε υπόψη μας ε, τις πραγματικότητες μεταξύ αυτών και το Brexit. Ε, και, ε, και πώς το βλέπετε δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Θα λειτουργήσει, γιατί όχι. Ωραία. Τα πάντα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και τούμπαλιν. Και φυσικά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ε, ομάδα παρακολουθήσεις που έχουμε στο κοινό. Ε, ευχαριστώ. Εισηγητή, ο κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία και να τα υπογραμμίσω. Θύμησε η Σάντρα ότι η συμφωνία αυτή είναι ε, πολιτικής σύνδεσης, οικονομικής συνεργασίας και εμπορικών συναλλαγών για απελευθέρωση των συναλλαγών στα θειακή. Γιατί το λέω αυτό γιατί κάποιο συνάδελφο μίλησε για ρήτρα δημοκρατική και βεβαίω υπάρχει ρήτρα δημοκρατία. Αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο τη συμφωνία και θα ήθελα να θυμίσω ότι είναι αμοιβαία η ρήτρα αυτή διμερής και απαιτητή και από τις δύο πλευρές. Και προφανώς η Γεωργία είναι ευαίσθητος τομέας. Ε, ε, προσωπεύει το 3,5% του ΟΕΠ παγκοσμίου ΑΕΠ θα έλεγα σχεδόν. Και είναι και ένας κλάδος προφανώς που θα πρέπει να προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να πω και ότι το υπόλοιπο 96,5% θα υποφεληθεί σαφώς από τη συμφωνία αυτή. Και το λέω γιατί μόλις το είπε η Σάντρα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα και έτσι επιθετικά στη Γεωργία, όπου βέβαια ο κύριος Χόγκαν, Επίτροπος Γεωργίας, έχει ένα πενιχρό ε, προϋπολογισμό 53 ε, δις το, το χρόνο 53 εκατομμυρίων για να αντισταθμίσει τις απώλειες. Το 2004 όταν σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις ήμασταν τότε 15 κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ποσόστοση σε τόνους από αυτό που συζητάμε σήμερα, που αναλογεί περίπου σε μισό χάμπουργκερ αναπολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με τις συμφωνίες με τον Καναδά, την Ιαπωνία κλπ. ανοίγουμε δυνατότητες, ευκαιρίες και αγορές για τους πολίτες μας. Θέλω να τελειώσω, Πρόεδρε, με δύο μηνύματα. Πρώτο, για τους φίλους και εταίρους μας της Μερκοσούρ. Θέλω να τους πω ότι πρέπει να βρούμε μια λογική λύση για το θέμα των αυτοκινήτων γιατί χωρίς αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τρόπο ικανοποιητικό. Επιστεύω ότι το θέμα των προσθεσμίων είναι βασικό για να βρούμε λύσεις. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να πω ότι πρέπει να είναι ευέλικτη, να προσπαθήσει να δει έτσι συνολικά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι δασμοί υπερβολικοί. Αν δούμε τι γίνεται σε άλλες συμφωνίες με άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά αν ανοίξουν οι συναλλαγές κατά 90-92% απελευθερωθούν, αυτό θα είναι προς όφελος και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τελικά, συνεπώς, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το γύρο των διαπραγματεύσεων και να αποδειχτούμε, όπως είπα και προηγουμένως, το ύψος των περιστάσεων. Τα θέματα τα υγειονομικά και φύτο υγειονομικά τα εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θύμησε η Σανδρά ότι θα πρέπει αυτά να γίνονται με αμοιβαιότητα. Έχουμε το πρόβλημα της Βραζιλίας, αλλά οι αρχές της χώρας αυτής το κατήγγελαν και ο αρμόδιος επίτροπος ε, το ανέλαβε πολύ γρήγορα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό ως πρόφαση για να μην προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για το σημείο 4 και θα πάμε στο σημείο 5 που είναι η προστασία ή η άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping και των επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό ήταν μία από τις επιτυχίες πεσινές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πιέσει το Συμβούλιο να συμφωνήσει για αυτή την νέα νομοθεσία. Θα θυμάστε ότι είχαμε τρία χρόνια που περιμέναμε την θέση του Κοινοβουλίου, τελικά τα καταφέραμε και μπορούμε με επιτυχία να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη ανάγνωση. Αποουσιάζει ο κύριος Φιέλνερ, και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ που τον αντικαθιστά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε ο Πρόεδρος Λάγκε, μιλώ εξ ονόματος του Κριστοφέρ Φιέλλερ, ο οποίος είναι εισηγητής για το θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Η, τα ε, συστήματα προστασίας ε, του εμπορίου είναι ένα από τα πιο λεπτά ζητήματα της εμπορικής πολιτικής κυρίως διότι υπάρχει μια διεθνώς αποδεκτή παρέκκληση από τους δασμούς ε, και χρεώνονται υψηλότεροι δασμοί από όσους μας δεσμεύουν στις συμφωνίες του ΠΟΕ και σε άλλες συμφωνίες. So, please, be quiet. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Thank you, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συμφωνίες για τον ε, ε, συγχρονισμό των ε, μέσων προστασίας του εμπορικού συστήματος είναι η πρώτη καινοτομία που γίνεται από το 1995 το τέλος του γύρου της Ουρουάης. Ματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου που ξεκίνησε το 2007 ε, ο τότε ο Επίτροπος Μάντελσον ε, έκανε μια πρόταση, υπήρχε και μια νομοθετική πρόταση από τον τότε Επίτροπο Ντεχούχτ. Και ε, τα μέσα γίνονται πιο προβλέψιμα, πιο διάφανα και πιο αποτελεσματικά με δύο λόγια, για να σταθώ στα πιο λεπτά ζητήματα και τι επέτυχε το Κοινοβούλιο κατά τη διαπραγμάτευσή του με το Συμβούλιο. Υπάρχει ο κανόνας για το χαμηλότερο δασμό. Ε, δεν θα ισχύει πλέον για δασμούς ε, ε, γενικότερα, αλλά κυρίως για ε, κανόνες κατά του ντάμπινγκ μόνο όταν έχουμε πάνω από το 17% του κόστου των αγαθών. Θα υπάρχει μία περίοδος τριών εβδομάδων πρώτερης κοινοποίηση ε, για να βεβαιωθούμε όμως ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν τρεις δικλείδες ασφαλείας και υπάρχει μια πρόταση ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους στασμούς. Θα έχουμε και ενδιαφερόμενα μέρη στην όλη διαδικασία τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύονται πλήρως από τι νέε διατάξεις σε και θα υπολογίζονται δασμοί βάσει του περιθωρίου και των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα υπάρχουν δασμοί για αγαθά τα οποία εισάγονται στην ε, ε, υπηρετική χώρα, εάν μπορούμε να αποφύγουμε τη ζημία για τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι ισορροπημένη έκθεση και ελπίζει να υπερψηφίσει η πλειοψηφία του των μελών και επίσης να προχωρήσουμε και την προκατακτική συμφωνία της Επιτροπής μας και να προχωρήσει και το θέμα στο Συμβούλιο. Ο κύριος Ντέιβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με τον Κρίστοφερ Φιέλνερ και την αξιολόγηση που κάνει και αυτά που μας διάβασε ο συνάδελφος. Είναι καλά νέα να έχουμε κάτι τέτοιο μετά από πέντε χρόνια. Μπορεί μακροπρόθεσμα να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη προστασία. Αν δούμε και σε τι κόσμο προχωράμε, αλλά καλό είναι που φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία και πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ ημών και του Συμβολίου και επομένω είναι καλό το γεγονό ότι φτάσαμε σε συμφωνία. Να ευχαριστήσω λοιπόν μέσω του κυρίου Βίνκλερ και του Κρίστοφερ γιατί ξέρω ότι ο Κρίστοφερ σε κάποια θέματα δεν ήταν καθόλου ενθουσιασμένο αλλά επέμεινε στη θέση του Κοινοβουλίου. Δύο ερωτήσει. Τη μία την αναφέρει και ο εισηγητής που είναι η θέση που αφορά την ε, ε Η Φαλοκρηπίδα Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τον εκτελεστικό κανονισμό, κατά πόσον θα υπάρχει ο εκτελεστικός κανονισμός σύντομα. Και το δεύτερο να αφορά το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με τον νέο κανονισμό, διότι υπάρχουν, ε, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, θα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα οι έρευνες όπως συμφωνήσαμε να γίνει νέα δουλειά για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων και να υπάρχουν και ε, κωδικοί για τους δασμούς, ε, να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Όλα αυτά είναι ε, σημαντικά καθήκοντα που απαιτούν πόρους και αν λειτουργήσει, πρέπει να λειτουργήσει το θέμα, πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα στον κανονισμό, αλλιώς θα είναι ανούσιος ο κανονισμός πολύ σύντομα μάλιστα. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή είναι ε, προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ο κύριος ε, Ζαντό για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον Ντέιβιντ και για τη δουλειά που έκανε ο εισηγητής. Δεν ήταν εύκολη αυτή η διαπραγμάτευση. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αρκετά στεναρή ε, τρόπον την διότι ε, βρεθήκαμε ενώπιον ενός συμβουλίου που για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του δεν επιθυμούσε και πολλά και ε, επέδειξε στεναρές αντιστάσεις στα περισσότερα σημεία Δυστυχώ. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή διότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε Σίγουρα δεν είναι επαναστατική, ιδιαίτερα στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά λαμβάνει υπόψη της αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ε, ε, ζητήματα, ακόμα και αν είναι στις πορυφές της προκατάληψης, αφορούν τις τιμές, ε, τις σχέσεις που πρέπει και τις εκθέσεις που πρέπει να ε, συντάσει και να δημοσιοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν όμως θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να συνειδητοποιήσουν απολύτως αυτό το οποίο επιτύχαμε, θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μέσα. Είτε όσον αφορά τη μεθοδολογία, αλλά και όσον αφορά τις δημοσίευσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχουμε ευρωεκλογέ του χρόνου και θα ήταν αδιανόητο να μην υπάρχει μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να ε, συνοψίζει τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και αυτά να αποτελούν βήμα της δημόσιας συζήτησης. Και να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μεν τέλεια, δεν επιτυγχάνουμε όλα αυτά που θέλουμε, ακόμα και εμείς οι οικολόγοι, αλλά πότε πότε καταφέρουμε να προχωρήσουμε κάποια πράγματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες. Η ερώτηση που είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς ε, ε, επειδή τώρα ασχολείστε με την νέα μεθοδολογία, και πώς θα φροντίσετε στις εκθέσεις σας να εντάξετε τα θέματα τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά και αν μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία για το τι θα κάνετε αυτά. Ευχαριστώ, Χέλμουτ Σόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους συναδέλφους, ευχαριστώντας και εγώ τον εισηγητή για τη συνεργασία του και για όλο αυτό το έργο, όλο αυτό το καιρό. Για όλη τη διαδικασία και πάντα ήταν δίκαιος και ε, ήθελε να συμπεριλάβει τα επιχειρήματά μας για να είναι και ισχυρή η θέση του Κοινοβουλίου. Καμιά φορά και ε, αντίθετα με τα δικά του πιστεύω ήταν αυτά που δεχόταν πραγματικά αξίεπαινος. Για το περιεχόμενο. Χαίρομαι πάρα πολύ και εκτιμώ για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο πρώτος ε, παγκόσμιος ε, πρωταγωνιστής που μιλάει για περιβαλλοντικό κόστος και κοινωνικό κόστος και το υπολογίζει κιόλας. Αν ακούτε τι, λένε ε, οι περιβαλλοντολόγοι, οι ειδικοί για το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα, θα μάθετε ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ και το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ ε, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί βαθύτατα. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ληφθεί αυτό υπόψη και να το θέσουμε υπόψη και των διεθνών εταίρων μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στα πολυμερή φόρα και ίσως κάποια μέρα στο μέλλον να έχουμε και ορισμό κοινωνικού ντάμπινγκ και περιβαλλοντικού και που μπορεί να το θεωρήσετε χρήσιμο. Εμείς το είχαμε προτείνει σε μια τροπολογία η οποία δυστυχώς απερίφθη. Και ορίζουμε ε, τι είναι το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και το κοινωνικό ντάμπινγκ και το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι όταν ρίχνουν τις τιμές ε, σε σχέση με τις ε, άλλες χώρες γιατί είναι πιο φτηνή η παραγωγή και είναι αθέμητη ε, πρακτική ανταγωνισμού. Και ιδιαίτερα όταν οι μέθοδοι ε, παραγωγής ε, χρησιμοποιούν κάποιες διαδικασίες που βλάπτουν το περιβάλλον και αυτό μειώνει το κόστος, να θεωρηθεί αυτό περιβαλλοντικό dumping. Λοιπόν, ποιος είναι ο δικός μας ρόλος να έχουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να προλαμβάνει και να αποτρέπει την κατάχρηση και των κοινωνικών προδιαγραφών και των περιβαλλοντικών. Και να φύγουν οι ορισμοί από τις αιτιολογικές σκέψεις και να μπουν στο κύριο κείμενο ε, και να το προωθήσουμε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τότε και μόνο τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα πρόοδου προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία Ζαμέ. Όλοι συμφωνούμε για την επιθετική πολιτική, την εμπορική της Κίνας ή τον προστατευτισμό του κύριου Τραμπ. Όλοι συμφωνούμε με αυτή την πυροβληματική θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Μια διαδικασία αντι-dumping, ναι, είναι κάτι ενδιαφέρον για αναγκαία μέτρα. Αλλά σε όλα αυτά τα μέτρα υπάρχει κάποια αφέλεια, θα έλεγα, θανατηφόρα μάλιστα. Οπότε μπορούμε να αναρωτηθούμε τι μέτρα ε, διαθέτει πραγματικά η Ευρώπη για να ερευνήσει για όλες αυτές τις χώρες. Εδώ βλέπω κάποια αδυναμία για το πώς ε, μπορούμε να μηνθούμε εμπορικά. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Μέτρα ή όχι, πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο μακριά από την Ευρώπη που προστατεύει και που θέλει να μας πουλήσει ο κύριος Γιούνκερ. Το κοινωνικό dumping γίνεται μέσα στην Ευρώπη. Οι αποσπασμένοι είναι κοινωνικό dumping. Πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Δεύτερον, για τους ρόλους του ΠΟΕ. Είμαστε οι μόνοι που τους στηρούμε. Ούτε η Κίνα τους θέλει, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες τους θέλει κανείς. Οπότε διαθέτουμε τα ίδια όπλα τελικά. Δεν νομίζω. Τέλος, χρειάζεται μια πολιτική υπέρ της κυριαρχίας, υπέρ των οικονομιών μας, υπέρ των ε, χωρών μας. Και το κείμενο αυτό δεν πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμάμαι κύριε Ζαντό τι είχατε πει που ήταν σωστό όταν μιλούσατε για μέτρα προστασίας ε, στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, σαφώς, εδώ προσπαθούμε να δούμε πώς θα προστατευτούμε από το dumping, δηλαδή πώς θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας εμείς. Με αυτά τα μέτρα το μόνο που κάνουν είναι ότι ζητάνε από τις χώρες ολόκληρου του κόσμου να μην προστατεύονται. Ε, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Ε, νομίζω ότι είναι εκ των προτέρων χαμένος αυτός ο αγώνας. Οπότε Όντω θα τη δώσετε αυτή τη μάχη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν πιστεύω ότι είναι η καλή λύση αυτή. Ο κύριος Μίλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί την Επιτροπή ΙΝΤΑ για την εξέταση του φακέλου αυτού. Εμείς, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, έχουμε δουλέψει σκληρά και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να είναι οικονομικά αποτελεσματικό, που είναι καλό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και γιατί ενσωματώνει και κοινωνικές αξίες στον μηχανισμό εμπορικής άμυνας. Και αυτό υπόθηκε και σήμερα το πρωί, είναι η πρώτη φορά που το καταφέραμε. σε ένα μέσο εμπορικής άμυνας. Τώρα για τις ερωτήσεις σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίζω με την ερώτηση του κύριου Μάρτιν. για την υφαλοκροπίδα συνεχίζεται η δουλειά στην ομάδα εμπειρογνωμόνων όπου προεδρεύει η Γενική Διεύθυνση Ταξούντ. Και θα λέγω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε συμφωνία. Και όταν ε, θα έχουμε δώσει απαντήσεις όλα τα τεχνικά ζητήματα, τότε θα ψηφιστεί στην ε, Επιτροπή για την ε, Εμπορική Άμυνα. Έχουμε πέντε διαφορετικά σχέδια και για το καθένα από αυτά είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε τελική λύση. Πάντως δεν μπορώ να προκαταβάλω βέβαια τα πράγματα. Δεύτερη ερώτηση. Για τους πόρους. Και είπατε ότι ο εξυγχρονισμός συμπεριλαμβάνει και κάποια νέα καθήκοντα. Είναι αλήθεια ότι ο εξυγχρονισμός αναθέτει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επί της ουσίας και κύρια, δεν πρόκειται για νέες αρμοδιότητες, πρόκειται για αλλαγή κανόνων. Για να εφαρμοστούν αυτοί πρέπει να καταρτιστούν οι συνάδελφοι για να είναι σε θέση να τους εφαρμόσουν τους νέους κανόνες και όχι τους παλιούς και άρα πρέπει να υπάρξει αυτή η ενημέρωση. Ακριβώς στα πλαίσια του εγχειρήματο αυτού ακολουθούμε νέες διαδικασίες ώστε να προχωρήσουμε σύντομα στην εφαρμογή των νέων αυτών κανόνων που συμφωνήθηκαν στο πακέτο εξυγχρονισμού. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν όταν αρχίσει τον επόμενο μήνα να ισχύει το νέο πακέτο, να είμαστε και εμείς έτοιμοι. Και επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να εργαστούμε με τους πόρους που διαθέτουμε, εφόσον βέβαια ο φόρτος εργασίας παραμείνει ως έχει σήμερα. Αν τότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Μία δυνατότητα είναι πάντα να υπάρξει κάποια μετάθεση. Αλλά όπως σας είπα, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με ό,τι έχουμε τώρα όσον αφορά τους ανθρωπίνους πόρους. Εφόσον δεν υπάρξει βέβαια επιπλέον φόρτος εργασίας που δεν προβλέπεται. Και υπάρχει και αρκετή ευελιξία ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες μας τις υποχρεώσεις. Περνάω τώρα στην ερώτηση του κύριου Σαντό. για το TGI, για τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές ε, και τα συνδικάτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει ενεργά το θέμα αυτό και θα το δείτε στην ανακοίνωσή μας, διάφορες ανακοινώσεις μάλλον, όταν σε αρχές του επόμενου μήνα αρχίσει να ισχύει ο εξυγχρονισμός. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στους κανόνες αυτούς και όπως συμφωνήσαμε στο πακέτο εξυγχρονισμού θα ενημερώσουμε για την εφαρμογή αυτών των νέων κανόνων. Οπότε μπορείτε να είσαστε ήσυχοι ότι θα το κάνουμε όπως πρέπει. Εμείς ε, θέλουμε όντω να συμπεριληφθούν οι προδιαγραφές και οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές, όπως έχει συμφωνηθεί εξάλλου. Τέλος, είπατε ότι δεν έχουμε αποτελεσματικά μέσα. Με κάθε σεβασμό διαφωνώ. Έχουμε ήδη αναλύσει την αποτελεσματικότητα των μέσων που διαθέτουμε στην αγορά. Ήδη στο παρελθόν, αν δείτε την αποτελεσματικότητα των μέτρων μας, θα διαπιστώσετε ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχή. Τα μέσα που έχουμε είτε για το dumping, είτε για επιδοτήσεις, με τον εξυγχρονισμό ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο αυτά τα μέσα, αυτά τα εργαλεία που έχουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικά είναι αποτελεσματικά και τα στοιχεία το δείχνουν αυτό ξεκάθαρα. Αυτά είχα να πω για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, Πρόεδρε. Και πάλι ευχαριστώ την Επιτροπή σας για το έργο της όσον αφορά το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την επικοδομητική σας στάση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Σεγητά, έχετε τίποτα να προσθέσετε. Ευχαριστώ πολύ και του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τα διαβιβάσω όλα αυτά τα συγχαρητήρια στον ίδιο τον εισηγητή. Εγώ απλώ τον εκπροσωπώ εδώ. Και από πλευρά του ΕΛΚ ένα σύντομο σχόλιο. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές ομάδες για ορισμένα θέματα. Ας πούμε, τη σημασία του κοινωνικού ντάμπινγκ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως έγινε πάρα πολλή δουλειά και συμφωνήσαμε γενικά και αξίζει η Επιτροπή μας να υποστηρίξει την τελική πρόταση. Ωραία. Άρα συνιστάτε να την εγκρίνουμε χωρίς άλλες τροπολογίες. Παρ' όλα αυτά θα σας πω μια προθεσμία. Σήμερα 6 ώρα λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, δεν περιμένω να κατατεθούν. Για να ψηφίσουμε με το καλό την άλλη φορά στην Ολομέλεια και να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή και θα είναι μεγάλη επιτυχία του Κοινοβουλίου. Επόμενο θέμα. Συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλούνται να εξέλθουν όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα δύο λεπτών.